Meine Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στην εδρία της Επιτροπής μας. Σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Βέσκοτ και την κυρία Μάστεν για θέματα που αφορούν την Αφρική και κυρίως το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Επίσης θα δούμε τον ε, αναπληρωτή πρόεδρο της Αλβανικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας και την ε, κυρία Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και εκπροσώπους της Αλβανικής Βουλής και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία. Ανακοινώσεις Προέδρου. Στις 8 Μαΐου η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είχε δεύτερη ανταλλαγή απόψε για τα θέματα του ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η συγκήτρια η κυρία είναι; Το Συμβούλιο επιθυμεί τον Ιούνιο να ορίσει τον πρώτο ειδικό εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και επειδή το ζήτημα είναι πήγον, θα σας παρακαλούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να ακολουθήσουμε τις προτάσεις του πρωτοτύπου και της τέταρτης αγγλικής ε, πρότασης. Προθεσμία κατάσταση απολογιών, αν θέλουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα, θα πρέπει να είναι η 16η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, έτσι ώστε στις 20 τέσσερις πλέον να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο όσο και κατεπήγον. Να περάσει και με ταχεία διαδικασία στην Ολομέλη. Εκτός εάν εγερθούν 40 μέλη και οργανώσουν μαζική αντίσταση. Θα ήθελα επίσης να σας πω συντομία ότι δεν πρόκειται να είμαι παρόν στη συζήτηση της δικής μου έκθεσης. Για ποιο λόγο. Στη Γερμανία έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα και δεν βοήθησε αυτό στις σχέσεις και στην ατμόσφαιρα μεταξύ μου και του κόμματός μου και δυστυχώς θα πρέπει να πάω πηγόντως για τη συνεδρία στο Προεδρείο του κόμματος. Καταλαβαίνετε όλοι οι πολιτικοί είστε ε, πώς έχει η κατάσταση. Σας έχω υποβάλει όμως την έκθεσή μου και θέλω να βάλω και λίγο ρυθμό. Να σας καλέσω λοιπόν μέχρι την άλλη Δευτέρα να καταθέσετε προφορικά ή και γραπτά τροπολογίες για να έχουμε την ευκαιρία την άλλη Δευτέρα στο Στρασβούργο νομίζω συνεδριάζει η Επιτροπή να το συζητήσουμε. Και αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, να ε, στείλω την ε, τελική εκδοχή για τις τροπολογίες. Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή? Για να μην καθυστερήσει η έκθεση, θα πρέπει να φροντίσουμε. Αν είχατε βοηθήσει όλοι μαζί να βγάλει καλύτερο αποτέλεσμα η Τσεντεού, δεν θα έπρεπε να φύγω σήμερα. Αλλά επειδή δεν το κάνατε, έχει η κατάσταση όσο έχει. Η κυρία Ντεκεζέρ έχει το λόγο. Βερονίκ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 Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, αλλά δυστυχώς στην πολιτική έχουμε και θλιβερές στιγμές, συχνά. Θα προεδρεύσει ο συνάδελφος κ. Κόβατσεφ. So, Γεια σας συνάδελφοι, σας καλωσορίζω και εγώ. Καλωσορίζω λοιπόν και τους προσκεκλημένους μας. με τους εκπροσώπους της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, όπως επίσης και τον υπεύθυνο για το τμήμα ε, Κεντρικής Αφρικής και Νοτιού Σουδάν να τους καλωσορίσω και τους δύο εδώ, και τον την κυρία Μάρσεν και τον κύριο Westcott, οι οποίοι θα συζητήσουν την προσπάθεια ειρήνευσης στο Βόρειο και στο Νότιο Σουδάν. Η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ε, εξωτερικής δράσης είναι σημαντική για το κοινοβούλιο μας. Ο κύριος Βέσκοτ θα μας ενημερώσει και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Αφρική και για τις ανησυχίες που έχουμε για την δημοκρατία του Κονγκό, το Μαλί και τη Γουινέα Μπισάου. Είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε και τις επενδυτικές δραστηριότητες στην Κεντρική Αφρική για να βοηθήσουμε έτσι στην ειρήνευση και την αποκατάσταση της ηρεμίας στην περιοχή. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην ειδική εκπρόσωπο του, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ή μάλλον πρώτα δίνω το λόγο στον κύριο Βέστχοτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στους συναδέλφους που ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι παρόν και γι' αυτό θα χρειαστεί να διαβρύνουμε λίγο τα θέματα προς συζήτηση σήμερα, έτσι ώστε τα μέλη που θέλουν περισσότερη ενημέρωση για την κεντρική Αφρική, τη δυτική Αφρική και την νότια μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Σήμερα συνεδριάζει συγγνώμη, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και για θέματα ανάπτυξης θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και γι' αυτό θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή των τελευταίων εξελίξεων στην κεντρική, δυτική και νότια Αφρική και μετά θα δώσω το λόγο στη Ρόζα Μάσντεν η οποία θα σας ενημερώσει για το Σουδάν και θα είμαστε στη διάθεσή σας σε λίγο χρόνο ε, για τις ερωτήσεις σας. Η κρίση στο κέρας της Αφρικής σας είναι γνωστή συνάδελφοι. Είναι μια κρίση η οποία έχει ξεσπάσει όμως και στη Δυτική Αφρική τους τελευταίους μήνες. Είναι κάτι το πρόσφατο και προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα ανταποκριθούμε, θα έλεγα, σε κάποιες καινούργιες καταστάσεις αναμαφέρομαι στο ε, Μπαλί και στην Γουινέα Μπισάο Όχι μόνο όμως αποκλειστικά σε αυτές τις χώρες. Η κατάσταση στο ΣΑΕΛ ήταν ε, εύθραυστη το, τους τελευταίους μήνες. Έχουμε συμφέροντα στην περιοχή, έχουμε εμπλακεί δυστυχώς και σε ε, παράνομο εμπόρεο ναρκωτικών, όπλων, απαγωγές υπηκών μας και γενικότερα απειλές. Έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική για το Σαχέλ, έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων πέρυσι σωστή στρατηγική και εύθετη, αλλά όχι χρονικά. Καθυστερήσαμε. Η ταχύτητα των εξελίξεων στο Σαχέλ και ειδικά στο Μαλί μας έδειξαν πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση και πώς η δράση την οποία προτείνουμε σήμερα ε, θα έπρεπε να είχε αναλυφθεί εδώ και δύο-τρία χρόνια για να αποφύγουμε τη σημερινή κατάσταση. Πάντως έτσι έχουν τα πράγματα και αυτό το οποίο προκλήθηκε από την εξέγευση, στην ανταρσία των στρατιωτικών στον Τάμασελ εδώ και ε, λίγους μήνες προκάλεσε προβλήματα, επιτάχυνε τις διαδικασίες, ιδιαίτερα στο βορρά του Μαλίου, όπου και οι Τουαρέγκ αυτονομιστές και οι τζιχαντιστές ουσιαστικά έχουν αναλάβει πλέον κάθε έλεγχο της περιοχής και η κεντρική κυβέρνηση του Μπαμακό δεν ελέγχει τίποτα στο βόρειο κομμάτι. Στο νότο τώρα του Μαλή ξέρετε ότι οδήγησε σε διάλυση των θεσμών και των τοπικών κυβερνήσεων. Η απάντηση της ΕΚΟΒΑΣ ήταν αρκετά γρήγορη θα έλεγα και ξεκάθαρη. Επέβαλαν αμέσως κυρώσεις έτσι ώστε να πισθεί η στρατιωτική χούντα να παραδώσει την εξουσία πίσω στην πολιτική μεταβατική κυβέρνηση και να οδηγήσει στις εκλογές οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τον μήνα Μάιο, αλλά τώρα πλέον έχουν αναβληθεί για μια, για ένα ευθετότερο, για μια ευθετότερη χρονική στιγμή. Η κατάσταση είναι προβληματική, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για τον ρόλο των στρατιωτικών και του λοχαγούς Σενάγκο, το ρόλο τους σε σχέση με τη μεταβατική κυβέρνηση της οποίας ηγείται ο τέος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Τραωρέ και ο ε, τέος πρωθυπουργός Διαρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά από τις συγκεκριμένες συνθήκες συνεχίζει να διακόπτει την βοήθειά της Εάν τυχόν υπάρξει συμφωνία για μια μεταβατική σταδιακή λύση και αν υπάρξουν αποδείξεις ότι θα ελέγχει την κατάσταση η πολιτική κυβέρνηση και όχι η στρατιωτική, τότε θα υποστηρίξουμε την πολιτική αυτή, την ενδιάμεση μετάβαση. Αν όμως ε, δεν υπάρξει ξεκάθαρη ε, επιθυμία επιστροφής της εξουσίας στις αρχές της πολιτικές, τότε θα δούμε αν πρέπει να εφαρμόσουμε το άρθρο 16 της Συνθήκης του Κοτονού, όπου θα σταματήσουμε να παρέχουμε βοήθεια μέσω της κυβέρνησης, μέχρι τη στιγμή που υπάρξει αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης. Η κατάσταση λοιπόν παρουσιάζει σημεία σύγχυσης, έχουμε κάνει θα έλεγα διαβήματα και προς την ΕΚΟΒΑΣ πήραμε μέρος στη συνάντηση κορυφής τους, παρακολουθήσαμε και είμαστε σε επαφή και με τις αρχές επιτόπου στον Παμάκο. Αν υπάρξει βέβαια απόφαση για συμφωνία στο Νότο, η κατάσταση στο Βορρά παραμένει ανησυχητική. Από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί η εξουσία της κυβέρνησης στην περιοχή αυτή με ειρηνικά μέσα. Η ΕΚΟΒΑΣ έχει ξεκινήσει μια διαπραγματευτική ε, ε, διαδικασία. Θα δούμε αν θα υπάρξει πρόοδος. Υπάρχουν όμως πολλές ε, ομάδες όπως η Αλκάιντα του Μαγκρέμπ που δεν έχουν καμία διάθεση να διαπραγματευτούν η αδίποτε λύση η οποία θα οδηγούσε στην εποκατάσταση του κράτους δικαίου στην περιοχή. Και έτσι μπορεί να αναγκαστούμε να ζητήσουμε στην, την προσφυγή στην βία για να αποκατασταθεί η πολιτική εξουσία στην περιοχή. Ε. Η ΕΚΟΒΑΣ έχει βοηθήσει και στρατιωτικά την κεντρική κυβέρνηση, αλλά περιμένουμε να υπάρξει ουσιαστική λύση στη διακυβέρνηση του Νότου και τότε θα δούμε τι θα γίνει. Λάβαμε ένα αίτημα από την ΕΚΟΒΑΣ να στηρίξουμε οικονομικά την μεταβατική δύναμη της ΕΚΟΒΑΣ η οποία αναμένει να παρέμβει εφόσον τη ζητηθεί από την κυβέρνηση του Μπαμακό. Δεν απαντήσαμε ακόμα, θα εξετάσουμε το αίτημα. Μπορούμε να απαντήσουμε μόνο στα πλαίσια των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και εφόσον ξεκαθαριστεί ποια είναι η κυβέρνηση με την οποία συνδιαλασσόμεθα και ποια θα είναι η εντολή αυτής της ενδιάμεσης σε αυτή τη φάση διαθέσιμη ε, στρατιωτικής δύναμης ΕΚΟΒΑΣ. Τώρα για τη Γουινέα Μπισάου η κατάσταση ε, έχει θα έλεγα σοβεί εδώ και πολύ καιρό και έχει και βαθύτερες ρίζες, πάρα πολλοί παράγοντες έχουν οδηγήσει σε αστάθεια τα τελευταία 30 χρόνια. Φιλετικές διαφορές, διαφορές ανάμεσα στους πολίτες και τους στρατιωτικούς, ισχυρή επιρροή από τους ε, λαθρεμπόρους ναρκωτικών, τρομερή διαφθορά. Ήδη έχουμε εφαρμόσει το 96 της συνθήκης του Κοτονού στις σχέσεις μας με τη Γουινέα Μπισάου. Είχε υπάρξει ελπίδα ότι η διαδικασία για την επιλογή Προέδρου η οποία είχε προχωρήσει, είχαμε περάσει τον πρώτο γύρο και περιμέναμε το δεύτερο, θα οδηγούσε σε μια κυβέρνηση η οποία θα είχε αρκετή νομιμοποίηση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μέσω της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας και των μεταρρυθμίσεων γενικότερα. Οι στρατιωτικοί φοβήθηκαν όμως μια τέτοια κυβέρνηση, διέκοψαν την διαδικασία, έκαναν πραξικόπημα και ε, εξεδίωξαν τους πολιτικούς εκτός από αυτούς που τους υποστήριζαν. δήλωσαν οι στρατιωτικοί ότι θα μεσολαβήσει ένας χρόνος για την επιστροφή σε μη στρατιωτικό καθεστώς και θα επιλέξουν αυτοί ποιο θα είναι το καθεστώς αυτό. Η ΕΚΟΒΑΣ δεν δέχτηκε αυτό την κατάσταση, ήδη πρότεινε να δημιουργηθεί και εκεί μια ενδιάμεση δύναμη η οποία να είναι διαθέσιμη 600 στρατιωτικών η οποία να βοηθήσει ε, να αποκατασταθεί η εκλογική διαδικασία. Η στρατιωτική κυβέρνηση δεν δέχτηκε την πρόταση ΕΚΟΒΑΣ και βρισκόμαστε τώρα πλέον σε αδιέξοδο. Υπάρχουν και στρατιωτικές δυνάμεις της Αγγόλα που παρέχουν τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση της, των δυνάμεων των τοπικών, των στρατιωτικών και αστυνομικών. Μισάγκ λέγεται η στρατιωτική αυτή αποστολή. Η ΕΚΟΒΑΣ είπε να αποσυρθεί η δύναμη αυτή, αλλά όταν μόνο οι δυνάμεις της ΕΚΟΒΑΣ αναπτυχθούν στην περιοχή και η κατάσταση παραμένει ασταθής, όπως είπα έχει διακοπεί η βοήθεια της Ευρωπαϊκής μέσω της εφαρμογής του 96 κοτονού. Η κατάσταση σε επίπεδο ανθρωπιστικό βέβαια στη χώρα δεν είναι τόσο κακή όσο στο Σαχέλ, γιατί στο Σαχέλ παράλληλα με την πολιτική κρίση έχουμε να βιώσουμε και μια βαθύτατα ανθρωπιστική κρίση. Ε, Παρ' όλα αυτά και στη Γουινέα Μπισάου η κατάσταση χειροτερεύει, δεν συλλέγονται πλέον οι νέες εσοδίες, κλείνουν οι τράπεζες, δεν υπάρχει ροή ρευστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως συνεχίζει να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της ΕΚΟ στο Σαχέλ, πέραν των ε, παρεμβάσεων μέσω των κυβερνήσεων. Πάντως και στις δύο αυτές χώρες η κατάσταση είναι ασταθής. Είμαστε σε στενή σχέση όχι μόνο με την ΕΚΟΒΑΣ αλλά και με τις άλλες χώρες της περιοχής, την Αλγερία, τη Μαυριτανία, και με άλλες χώρες οι οποίες ε, ε, είναι γειτονικέ, συνεργαζόμαστε και με τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα για τις άλλες χώρες όπου οι εξελίξεις ήταν λίγο καλύτερες. Το Μαλάβι την περίοδο του Πάσχα υπήρξε μια κρίση μετά από τον αδόκητο ε, θάνατο του βασιλέως Μουτεφίκα ε, το Σύνταγμα προβλέπει την αντικατάστασή του από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος θα αναλάβει την Προεδρία της χώρας, αλλά ορισμένοι από τους υποσταρικτές του κυρίου Μουφερίκα δεν ήσαν υπέρ μιας τέτοιας αντικατάστασης, γιατί η Τζόις Μπάντα δεν είχε καλές σχέσεις με τον βασιλέα Μουφερίκα και είχε εκδιωχθεί η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με την χώρα της Νοτιού Αφρικής και με τη σωστή θέση ε, των ενόπλων δυνάμεων του Μαλάουι που είχαν πει ότι θα στηρίξουν ε, τη συνταγματική λύση οδήγησε σε μία θα έλεγα ήρεμη συνταγματική θα έλεγα επίλυση του προβλήματος. Τώρα πρόεδρος είναι η κυρία Τζόις Μπάντα. Απεφεύχθη η συνταγματική κρίση και έτσι αποφύγαμε να επαναλάβουμε αυτά τα οποία είχαμε βιώσει στο παρελθόν. Τώρα μετά από αυτό το Μαλάουι για τη Ζιμπάμπουε και μετά από την απόφαση για απόσυρση ορισμένων από τα περιοριστικά μέτρα εμείς ε, δημιουργήσαμε την Επιτροπή Υπουργικής Επανεμπλοκής, επαφή δηλαδή με, τις, ε, με τα τρία μεγάλα κόμματα. Ε, έγινε μια πρώτη επαφή στις Βρυξέλλες, συμφωνήσαμε για μία θα έλεγα πορεία προς το μέλλον επί τη βάση 96 μέτρων που υιοθετήθηκαν τον προηγούμενο Ιούλιο και θεωρούμε ότι έχει υπάρξει αρκετή πρόοδο σε σχέση με την εφαρμογή του νέου συντάγματος και τις <coughs> εκλογές που προβλέπονται για το επόμενο έτος. Και θα δούμε αν έχουν υπάρξει βήματα πρόοδου έτσι ώστε να μειώσουμε τις κυρώσεις. Έχουμε λοιπόν ε, μια μορφή θετικού διαλόγου με τις εμπλεκόμενες εκεί πολιτικές δυνάμεις. Τέλος θα αναφερθώ στην δημοκρατία του Κονγκό. Έχει ήδη, θα έλεγα, ε, υπάρξει μια νέα κυβέρνηση μετά από τις τελευταίες εκλογές. Είναι τεχνοκρατική κυβέρνηση, είναι ενθαρρυντικό, γιατί τώρα έχουμε συνομιλητές και μπορούμε να εξετάσουμε την με πιο αποτελεσματικό τρόπο χορήγησης της κοινοτικής βοήθειας προς τη χώρα αυτή όπου ένας από τους θέους στρατιωτικούς ε, εξεγερμένους ηγέτες επέστρεψε στις, ε, ε, είχε επιστρέψει στο στρατό, τώρα όμως αναχώρησε εκ νέου και υπάρχει θα έλεγα μια σύγκρουση ουσιαστικά ανάμεσα στις επίσημες ένοπλες δυνάμεις και τους τασιαστές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Για το Σουδάν θα σας τα πει η Ρόζα Λίντα η κατάσταση εκεί έχει χειροτερεύσει τις τελευταίες εβδομάδες δραματικά. Υπήρξε και η εισβολή προς την πόλη στον οικισμό του Χέτζλικ από δυνάμεις του Νοτιού Σουδάν. Εμπλεκόμεθα στις, ε, στην διαφορά αυτή μαζί με άλλες ε, διεθνείς ε, δυνάμεις εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας είναι πολύ σημαντικό η ομοφωνία της διεθνούς κοινότητας να συνεχιστεί έτσι ώστε η πίεση και προς τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μια ανακοχή, να επιστρέψουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και έτσι και ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας και το Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν ε, καταλήξει σε κοινέ θέσεις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 Ε, President ε, για τις ε, βίες εκεί συγκρούσεις και μάλιστα ζητήθηκε αποχώρηση των δυνάμεων από το Χέικλικ. Βέβαια έγιναν καταγγελίες για την κλιμάκωση το, της βιότητας και τον βομβαρδισμό των διαμερισμάτων του Νοτίου Σουδάν. Συζητήθηκε στις 23 Απριλίου το ζήτημα του Βορείου και Νοτιού Σουδάν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Μέχρι τότε απέσυρε το Νότιο Σουδάν τις δυνάμεις από το Χέζλικ και απευθύνθηκε έκκληση και στις του Βορείου και του Νοτιού Σουδάν να ε, σταματήσουν τις εχθροπραξίες είτε άμεσα είτε έμεσα, να αποσύρουν το προσωπικό ασφαλείας από την περιοχή ABA και να αποφύγουν οποιασδήποτε προκλητικές ενέργειες, ε, ακόμη και ε, μισαλόδοξες δηλώσεις. Επίσης, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και τη, του πάνελ υψηλού επίπεδου για την εφαρμογή των συμφωνιών σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνεί διεθνείς εταίρους προκειμένου να εξασφαλιστεί και οι δύο κυβερνήσεις θα πραγματοποιήσουν τα απαραίτητα διαβήματα και τα βήματα, τα στάδια που πρότεινε το Συμβούλιο. Ε, στις 24 Απριλίου το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, της ε, Αφρικανικής Ένωσης κατήρτισε έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα βήματα για την κατάπαυση των εχθροπραξιών και την επαναφορά και των δύο πλευρών στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και αυτός ο οδικός χάρτης στη συνέχεια επιδοκιμάστηκε και από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα 2046 της 27 Μαΐου. Και μάλιστα και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσόρισε θερμά αυτό το ψήφισμα. Θεωρούμε ότι η αμόφωνη ε, έγκριση του ψηφίσματος του κεφαλαίου 7 ήταν ένα σημαντικό, μια σημαντική διπλωματική επιτυχία και ένα καλό παράδειγμα στενής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης. Και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουμε πια μια διεθνή συνένεση για το τι μέλη γενέστε και τι ιδέωνει. Είναι το να από εδώ και πέρα. Φυσικά το χρονοδιάγραμμα είναι σχετικά φιλόδοξο και περιέχει ε, αυστηρά κριτήρια ενημέρωσης και για, και για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και για το Συμβούλιο Ασφάλειας και Ειρήνης της Αφρικανικής Ένωσης και υπάρχει και απειλή ε, κυρώσεων μη στρατιωτικών από το, από το Συμβούλιο Ασφαλείας με βάση το άρθρο 41 αν οποιαδήποτε από τις πλευρές δεν ε, συμμορφωθούν με τον οδικό χάρτη. Τώρα, βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κρατήσει αμύωτη την πίεση και στι διακυβερνήσει για την εφαρμογή του ψηφίσματο χωρί αλλαγέ και χωρί καθυστέρηση. Και μάλιστα είχαμε και τη δήλωση της Υπατής προσώπου της 5 η Μαΐου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τον πρόεδρο Μπέκη και ε, τον πρόεδρο Μίλες καθώς και τον ειδικό επιστελμένο του ΟΗΕ, του Χαϊλέ Μενκέριος. Και θα γίνω συζητήσει με τις δύο πλευρές. Είχαμε στενές επαφές και με πολύ σημαντικούς περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, Κίνα, Αιθιοπία, Αίγυπτο, Νότιο Αφρική, Τουρκία και πολλές ε, άλλες χώρες. Επιπλέον συναντηθήκαμε με ειδικού επιστελμένου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Νορβηγία. Οι κυβερνήσει του Βορείου και Νοτιού Σουδάν δέχτηκαν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλεία και συμφώνησαν να καταπαύσουν τι εχθροπραξίε. Είναι σημαντικό όμω οι δηλώσει να συνοδευτούν και από έργα και την άμεση επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Ευελπιστούμε ότι ε, στο μέλλον το πάνελ θα θα συγκαλέσει ε, συνάντηση στην Αντισαμπέμπα του Μηχανισμού Ασφάλειας και Προστασίας προκειμένου να καλυφθούν ε, οι ανησυχίες περί ασφάλειας και των δύο πλευρών. Άλλο σημαντικό θέμα είναι να κινητοποιηθεί ο κοινό μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευση ελέγχου των συνόρων που καταρχήν έχει συμφωνηθεί από, από τις εμπλεκόμενες πλευρές σε συμφωνία με τους διεθνείς παρατηρητές με συμμετοχή παρατηρητών από Βόρειο και Νότιο Σουδάν. Ο μηχανισμός αυτός θα εξασφαλίσει την ε, έμπρακτη εφαρμογή της κατάπαυσης των εχθροπραξιών στα σύνορα. Χαιρόμαστε γιατί πριν από δύο μέρες επιβεβαιώθηκε η αποχώρηση όλου του αστυνομικού προσωπικού του Νοτιού Σουδάν από, την περιοχή ABA και ελπίζουμε ότι και το Βόρειο Σουδάν με βάση το ψήφισμα 2046 θα πράξει κάτι αντίστοιχο. Οι τάσεις πάντως μεταξύ Βορείου και Νοτίου Σουδάν σχετίζονται με την ε, κατάσταση στο κράτος ε, Blue Nile. Εκεί δεν έχουν σταματήσει εχθροπραξίες δυστυχώς και οι συγκρούσεις μεταξύ του SPLM ε, και των, του, επαναστατικού, του επαναστατικού κινήματος του Σουδάν και των δυνάμεων του Σουδάν συνεχίζονται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να καταλήξουμε σε πολιτική λύση για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση και χαιρόμαστε που το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας προβλέπει ότι και ε, το SPLM North και η κυβέρνηση του Σουδάν θα πρέπει να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Μπέκη και τον ε, Πρωθυπουργό Μελές προκειμένου να καταλήξουν σε συνενετική λύση με βάση τη συμφωνία πλαίσιο που έχουν ε, προσυπογράψει στις 26, 28 Ιουνίου πέρυσι και οι δύο πλευρές. Επίσης, ε, λυπόμαστε που η κυβέρνηση του Σουδάν δεν έχει δεχτεί ακόμη την τριμερή πρόταση για την ε, πρόσβαση των ε, ανθρωπιστικών δυνάμεων στο, στον άμαχο πληθυσμό του Blue Nile που έχει υποβληθεί από τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ και βρίσκεται υποσυζήτηση ήδη από το Φεβρουάριο. Ω ε, διάμεσο βήμα ζητούμε από την κυβέρνηση του Σουδάν να επιτρέψει πρόσβαση τη ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον άμαχο πληθυσμό σε περιοχέ που μαστίζονται από τι συγκρούσει ε, στι δύο αυτέ πολιτείε. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί τα μάλλα για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βόρειο και Νότιο Σουδάν. Στο Νότιο Σουδάν έχουμε προβληματισμό μετά από ε, εκθέσεις για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το SPLA. Και ο ύπατο αρμοστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ναβι Πίλεϊ, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σουδάν μετά από άνοιγμα της κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν και ελπίζουμε ότι και η κυβέρνηση του Σιδάν θα προσκαλέσει την υποταρμοστή να επισκεφθεί το Χαρτούν. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Σουδάν, συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε από τη φυλάκιση αντιφρονούντων δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και ειρηνικών, διαδηλωτών φοιτητών είχαμε μια δημοκρατική κυβέρνηση που είπαμε ότι θα, σέβεται τη διαφορετικότητα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Θέλουμε λοιπόν να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και να έχουμε μια πραγματικά περιεκτική κυβέρνηση, δημοκρατική και στις δύο χώρες, το Βόρειο και το Νότιο Σουδάν. Μείναμε ικανοποιημένοι από την επίσκεψη του Πρόεδρου το Μάρτιο στις Βρυξέλλες. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι η κυβέρνηση ε, θέλει να προσχωρήσει στη Συμφωνία του Κοτονού και πιστεύουμε ότι το Κοτονού θα αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη βάση για ανάπτυξη των σχέσεων με τον Νότιο Σουδάν και για τη δημιουργία διαλόγου για ζητήματα που αποτελούν τον πυρήνα αυτή τη εταιρική σχέση, τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλο, και παρόλο που η διεθνή προσοχή επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή κυρίω στι σχέσει μεταξύ Βορείου και Νοτιού Σουδάν, εξαιτία του δικού χάρτη και του ψηφίσματο του Συμβουλίου Ασφαλεία στο ΙΕ, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε και την κατάσταση στον Ταρφούρ. Η κατάσταση ασφάλειας στον Ταρφούρ ε, έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να μην είναι καλή. Ε, έχουμε με πολλές ε, ενέργειες εγκληματικές, σημαντικά επεισόδια καταπάτης ασφάλειας στο νότιο Νταρφούρ. Θεωρούμε ότι ακόμη δεν υπάρχει πρόσβαση στο Τζάμπλναρ και η UNAMID εξακολουθεί να έχει περιορισμένη ελευθερία κινήσεων η παρουσία 1,7 εκατομμυρίων εσωτερικά εκτοπισθέντων σε καταβλισμούς δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση του Σουδάν και το κίνημα ισότητα, απελευθέρωση και δικαιοσύνη να εφαρμόσει το, την ειρηνευτική συμφωνία που υπέγραψαν τον προηγούμενο Ιούλιο και να ε, να, εφαρμοσ... να, να αναλάβει μια διοίκηση στον Ταρφούρ που θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία. Δυστυχώ δεν είχαμε σημαντική πρόοδο του τελευταίου μήνε. Η κυβέρνηση του Σουδάν δυστυχώ δεν ε, τήρησε τι οικονομικέ υποχρεώσει που είχε αναλάβει και η κατάσταση ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο τη προσοχή μα. Ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ κύριε Μάστον και κύριε Βέσκο που μας δώσατε αυτή την πληροφόρηση ε, από τα μέσα ε, για την Αφρική και ιδιαίτερα το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Ντεκεζέρ. Είναι επίσης επικεφαλής της αντιπροσωπείας παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των ε, καταστάσεων στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση στον κύριο ότι θέλω να κάνω σχετικά με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Μας είπατε δύο λόγια για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, αλλά είχα την αίσθηση ότι ήταν σχετικά αισιόδοξα αυτά που μας λέγατε. Εντάξει, συμφωνώ. Σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι το Μαλί, η Γουινέα, Μπισάου, ε, συχνά σε καταστροφικές καταστάσεις, η κατάσταση λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό βεβαίως είναι λιγότερο κρίσιμη, σοβαρή. Ωστόσο, Ε, ε, μιλάτε για μια κυβέρνηση που επιτέλους έχει εκλεγεί και τα λοιπά και ξαναρχίζει τη συνεργασία. Θα ήθελα να θυμίσω όμως ότι είχαμε πάει ε, με την κυρία Νετέλτσεβα για την παρακολούθηση των εκλογών και καθόλου δεν εγκρίναμε τις εκλογές ως προς τη διεξαγωγή τους. Υπήρχαν συμπτώματα νοθείας και σε ό,τι αφορά τους ακτιβιστές ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα στρατοδικείο έκανε μια ε, δίκη, που, ε, εντάξει ήταν δίκαιη δίκη, αλλά τι γίνεται με αυτούς που θεωρούνται δολοφόνοι. Είναι πλήρης η ατιμορρησία, είναι ελεύθερη και δεν έχει γίνει ακόμα ακουστή η έκκληση της κυρίας Σεβαγιά και άλλες δολοφονίες ακόμα δεν έχουν εξηχνιαστεί. Η κατάσταση δεν παραμένει άκρος, άκρος ανησυχητική σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάξει, εγώ λέγω ότι ε, αν ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επαναλαμβάνει τις συνομιλίες και τη βοήθεια και τις σχέσεις με τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, καλώς πράττει, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να συνδέεται αυτό με κάποιους όρους, με τη ε, σημαντική βελτίωση στον τομέα αυτό. Και εμείς, τουλάχιστον η πολιτική μου ομάδα και ελπίζω και οι υπόλοιπε, θα καταθέσουμε ένα κατεπήγον. Απευθύνω μια έκκληση προς άλλες πολιτικές ομάδες να κάνουμε ένα κατεπήγο για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό που θα σας θυμίζει ευλόγως τα σημεία τα οποία θέλουμε να δούμε πρόοδο στη χώρα αυτή. Κυρία Μάρστερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισκόπηση που μας δώσατε της κατάστασης στο Σουδάν και ιδιαίτερα στο Νότιο Σουδάν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω Όταν σήμερα κάνετε την ανάλυση σας, και χαίρομαι βεβαίως που υπάρχει ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με οδικό χάρτη, με χρονοδιάγραμμα, επι, επιτέλους θα έλεγα. Αλλά αν δω πώς είχε κατάσταση πέρυσι τέτοιο καιρό, σε σχέση με τη σημερινή, ο οποίο όλα τα προβλήματα που δεν είχαν λυθεί, είτε είναι τα θέματα της ηθαγένειας, ή πώς θα μοιράσουν το πετρέλαιο, ή τα θέματα των συνόρων, εκκρεμούν στο ακέραιο ακόμα. Και σχεδόν εμπόλεμη σύρεξη μεταξύ των δύο χωρών, οι βομβαρδισμοί στο γαλάζιο νήλο και όλα αυτά τα προβλήματα να φτάσει η ανθρωπιστική των δυο χωρων οι βομβαρδισμοι στο γαλαζιο νειλο και ολα αυτα τα προβληματα να φτασει η ανθρωπιστικη βοηθεια ο όλο και πιο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η Κίνα που φέρεται τώρα ως διαμεσολαβητής και ε, καταθέτει στο τραπέζι δισεκατομμύρια δολάρια όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο ε, δεν είναι και επιτυχία. Δεν ήμασταν αρκετά ε, εκεί οξυδερκείς, ε, προσεκτικοί, επίμονοι Ποια είναι η ανάλυση σας, κυρία Μάρστεν, σε σχέση με αυτό το έτος που ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν και τι αμέλησε να κάνει, δεν έπραξε σωστά η διεθνής κοινότητα επιβάλαμε την ανεξαρτησία της χώρας αυτής και εγώ είμαι η πρώτη που θα πω ότι ήταν απαραίτητο για να αποφευχθεί ο πόλεμος. Ε, αλλά εάν ε, με αυτή την ανεξαρτησία και πάλι δεν αποφεύγουμε τον πόλεμο, τίθενται κάποια ερωτηματικά. Και ιδιαίτερα για το ρόλο της Κίνας και το θέμα του πετρελαίου και του δεχομένου αγωγού που θα περνάει μέσα από την Κένια. Μεγάλη υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεκεζέρ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, και εμείς θεωρούμε ότι το ψήφισμα το ομόφωνο του Συμβουλίου Ασφαλείας της ε, Δευτέρας Μαΐου ε, δείχνει τον οδικό χάρτη μετά την απόφαση 24 Απριλίου του αντίστοιχου οργάνου της ε, Αφρικανικής Ένωσης οι όροι είναι σαφείς, να σταματήσουν οι ε, συμπεριλαμβανομένων και των ε, βομβαρδισμών. Τα θέματα ε, τα ανέφερε και η κυρία Ντεκεζέ στην τοποθέτησή της, ιδιαίτερα το πετρέλαιο. Η χάραξη των συνόρων, που είναι πάρα πολύ περίπλοκη, με μεθόριος πάνω από χίλια χιλιόμετρα. Τι γίνεται με την ηθαγένεια των πολιτών ε, της κάθε μιας από τις δύο χώρες και επίσης πώς θα μπορεί να φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Στα πλαίσια αυτά παρατηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία την επιστράτευση και στις δύο χώρες και επίκειται πόλεμος από ό,τι φαίνεται. Και θα ε, ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας και των δύο ως προς τη δυνατότητα κινητοποίησης και ε, παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Πιστεύω ότι το θέμα του πετρελαίου είναι ουσιαστικό. Γνωρίζουμε ότι είναι αναγκασμένο το Νότιο Σουδάν να εξαγάγει αυτή την πρώτη ύλη ε, διαμέσου του Σουδάν και των λιμανιών του στο βορρά και τις ε, καταχρήσεις που γίνονται και τις εξωφρενικές τιμές που πρέπει να καταβάλουν. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Μάρστεν και να τη ρωτήσω ε, πώς θα γίνει η ένταξη του Νοτιού Σουδάν ε, στη Σύμβαση του Κοτονού είναι οι χώρες ΑΚΕ που συμμετέχουν εκεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί σαφή κριτήρια και υποχρεώσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και γίνεται και ειδική αναφορά στο σεβασμό ε, της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του Σουδάν έχει προσαχθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. και Θα πρέπει να ε, λογοδοτήσει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αρχές του Νοτίου Σουδάν θα υποβάλουν αίτηση ένταξη στις χώρες ΑΚΕ, στη Σύμβαση Κοτονού ή θεωρούν ότι αυτό θα είναι ένα επιπλέον στοιχείο που θα περιπλέξει τις σχέσεις του με το Σουδάν που είναι ήδη πάρα πολύ περίπλοκες και δύσκολες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you, Mrs. Now the floor. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Κυρία Γκόμες που είναι επίσης επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας παρακολούθηση των εκλογών στο Σουδάν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία αυτή, πριν φύγει ο κύριος Γουέσκοτ, ε, για να το ρωτήσω κάτι για μια χώρα που καλύπτουν ε, πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η δεύτερη σε σημασία και ε, η έδρα της Αφρικανικής Ένωσης, η Αιθιοπία. Ένας ε, δημοσιογράφος ε, που είναι στη φυλακή στην Αιθιοπία βραβεύτηκε πρόσφατα με το βραβείο Pen Award και επίσης άλλοι δημοσιογράφοι διώκονται και φυλακίζονται. Και θα ήθελα να σας πω ότι τα όσα συμβαίνουν στην Αφρική και ιδιαίτερα στη Δυτική Αφρική συμβαίνουν απουσία και ρήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεράστιε οι συνέπειες της οικονομικής, πολιτικής και χρηματοοικονομικής κρίση στην Ένωση. Και αυτό ανακλάται και στην εξωτερική μας πολιτική. Βεβαίω όλα αυτά είναι πολύ πέραν του ε, πεδίου αρμοδιοτήτων σα. Αλλά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση προβληματίζεται, το σκέφτεται Ήταν σφάλμα η κατάργηση της αποστολής ΕΠΑ που είχαμε ε, στην ε, Γουινέα Μπισάου. Όταν έχει μεταρρύθμιση ε, του τομέα ασφαλείας, δεν ξέρω ποια ήταν η πρόφαση. Δεν είναι η περίπτωση αυτή που χρειαζόμαστε να φύγουμε, να είμαστε απόντες. Χρειάζεται να συμμετέχουμε περισσότερο εκεί και όχι λιγότερο. Και συμφωνείτε μαζί μου ότι πέρα από τα όσα μας είπατε για το τι συμβαίνει στο Μαλί, στη Γουνέα Μπισάου και πώς συνδέονται όλα αυτά και πώς ε, αναπτύσσονται τα εγκληματικά ε, δίκτυα και συνδέονται με την Αλκάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέπ. Μήπως βλέπετε ε, στη Γουνέα Βισάου να διεξάγεται ένας πόλεμος μεταξύ Νιγηρίας και Αγγόλας Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι την κυρία Μάρσεν και χαίρομαι που είναι οποίο μας και μας ενημέρωσε. Βλέπετε καμία πρόοδο ε, στο νότιο Σουδάν ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας είπατε ότι ε, έχει προσκληθεί, είπατε, ε, εκπρόσωπος και ελπίζω να έρθει. Ή μήπως ο πόλεμος είναι μια δικαιολογία για να μην έχουν καμία πρόοδο. Και θέλω να σχολιάσετε και κάτι που διάβασα στους New York Times, που έλεγε «Δώστε μια ευκαιρία στον πόλεμο» ο τίτλος. Και αναφερόταν ε, στα τακτενόματα μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν. Και εννοούσε το δημοσίευμα ότι είναι ένας τρόπος αυτός να απομακρυνθεί από την εξουσία ο κύριος Μπασίρ γιατί δεν έχει επιτευχθεί καμία πρόοδος και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Ευχαριστώ κύριος Τάνοκ που είναι και εισηγητής για το κέρας της Αφρικής. Και μετά θα παρακαλούσα να απαντήσετε. Uh, Καλώς ορίζω την Ντέιμ Ρόζαλιν και τον Νίκ. Προφανώς ενημερώσατε για το Σαχέλ, γιατί εγώ μπήκα καθυστερημένα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πολλά λιβικά όπλα χρηματοδοτούμενα από Κατάρα από ό,τι φαίνεται καταλήγουν στα χέρια της ε, Ισλαμικής Αλκάιντα του Μαγκρέμπ και που συνεργάζονται από ό,τι φαίνεται με τους αυτονομιστές ε, της περιοχής. Η περιοχή αυτή μπορεί να υποστηρίξει την αυτονομία της ή μήπως θα δούμε να δημιουργείται μια νέα Σομαλία παράδεισο για όλους τους τρομοχράτες τζιχαδιστές και απειλή για το σύνολο της περιοχής. Μήπως είμαι πολύ απεσιόδοξος. Ένα άλλο θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ή την επιτροπή μας, αλλά επηρεάζει την Αφρική. Δεν είμαι στην αρμόδια επιτροπή, αλλά φαίνεται ότι προσπαθεί να δημιουργήσει νέους κανόνες για τις πιθανές πληρωμές προς τις κυβερνήσεις από τις επιχειρήσεις εξορρυκτικών δραστηριοτήτων, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πολλά εμπορικά προβλήματα, αλλά θα ανοίξει επίσης και τις θύρες στην κυριαρχία των Κινέζων, γιατί οι Κινέζοι δεν ασχολούνται και πάρα πολύ με τέτοιου είδους λεπτομέρειες πόσο μπορούμε εμείς ε, να ε, είμαστε θα έλεγα στο ίδιο επίπεδο με τους Αμερικανούς σε σχέση με την διαφάνεια και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα για την Ντέιμ Ρόζαλιν για τον Νότιο Σουδάν. Άκουσα κάπου ότι έχουν λίγα ε, χρήματα σε συνάλλαγμα γιατί φαίνεται δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πετρέλαιο που να βγαίνει από τον Νότο και ο Νότος δεν θα έχει καθόλου έσοδα σε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, αν τελειώσουν τα χρήματα στο Νότιο Σουδάν θα δημιουργηθεί μια σοβαρή οικονομική κρίση και αυτό θα περιπλέξει τις στρατιωτικές συγκρούσεις οι οποίες σοβούν ήδη. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους φιλοξενούμενους για να δώσουν τον πρώτο γύρο απαντήσεων. Ερώτηση της κυρίας Κάιζερ για το Κογκό. Είναι πολύ εύθραυστη χώρα και πολύ εύθραυστη περιοχή των μεγάλων λιμνών. και είδαμε ότι ο ηγέτης στασιαστής Μπάντα εγκατέλειψε για μια ακόμη φορά τις στρατιωτικές επίσημες δυνάμεις και στασίασε. Και αυτό επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητα της περιοχής. Εμείς είδαμε τις, τα, τα συμπεράσματα από την εκλογική διαδικασία η οποία παρακολουθήθηκε, διαβάσαμε προσεκτικά τα συμπεράσματα και καταλήγουμε στο ότι πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα προς την κατεύθυνση αυτή και πρέπει να υπάρξει αυτή η μεταρρύθμιση πριν τις επόμενες εκλογές. Μπορούμε να βοηθήσουμε για να γίνει αυτή η αλλαγή. Απαιτείται ο συνδυασμός των μέσων μας με τις δικές τους επιθυμίες. Δεύτερον, η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκατάσταση κράτους δικαίου, τάξης, νόμου, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη χώρα μέσω των δύο αποστολών ΚΕΠΑ για την αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση των δυνάμεων καταστολής, των δυνάμεων της τάξης μάλλον της περιοχής κάτι το οποίο επηρεάζει την τήρηση της τάξης για το σύνολο της χώρας, όπου εκεί οι πληθυσμοί, ιδιαίτερα στο ανατολικό κομμάτι, είναι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους καταχρήσεις. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο Καμπιλά, όταν μπορέσω να τον επισκεφθώ εγώ, είτε ο Επίτροπος Πιμπαλσκ. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε λοιπόν τις εργασίες των διαφόρων οργανώσεων που προσπαθούν να βελτιώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί όπως και στο παρελθόν. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα μείωση ένδυας επιμέρους τα οποία πρέπει να συνεχιστούν. Τώρα για την Αιθιοπία. Και εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κάτι που δεν αγνοούμε συνεχίζουμε να βοηθάμε αναπτυξιακά τη χώρα σε υψηλό επίπεδο, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ένα κρίσιμο πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση. Υπογραμμίζουμε πάντα την σημασία του να υπάρξει πολιτικός χώρος για το άκουσμα και εναλλακτικών πολιτικών σκέψεων και ήμασταν αρκετά ικανοί γιατί συνεχίζουμε θα έλεγα να ενισχύουμε και την κοινωνία των πολιτών και πάντα φέρνουμε στην επικαιρότητα θέματα για θα έλεγα την απελευθέρωση ορισμένων που είχαν συλληφθεί καταχρηστικά. Συνεργαζόμαστε με τη Σουηδική κυβέρνηση και για την περίπτωση των κρατουμένων Σουηδών δημοσιογράφων μια κατάσταση η οποία θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να ξεπεραστεί αλλά δεν θα ξεχαστεί. Για τη Δυτική Αφρική είπατε πολύ σωστά ότι είχαμε μια αποστολή και πά ε, στο Ιγουνέα Μπισάου η οποία έχει λήξει. Στη Γουινέα Μπισάου ε, το θέμα είναι αν θα πιστέψουμε αυτά που μας λένε για τις μεταρρυθμίσεις ή αν θα πιστέψουμε αυτά τα οποία βλέπουμε γιατί δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν και πολύ. Τα τελευταία γεγονότα δείχνουν ότι μόνο τα μάτια μας μας λένε την αλήθεια. Βέβαια υπήρξε μια προσπάθεια όταν τα στρατεύματα της Αγκόλας θα μπορούσαν να παίξουν καλύτερα τον ρόλο αυτό γιατί ομιλούν την πορτοκαλική, αλλά απέτυχαν. Τώρα το αν θα πετύχει μια δύναμη της ΕΚΟΒΑΣ καλύτερα από τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, εμείς είχαμε ένα ειλικρινέστατο διάλογο με την ΕΚΟΒΑΣ. Τους είπαμε ότι αν μπείτε θα υπάρξει λύση μόνο αν φύγουν οι στρατιωτικοί από την πολιτική, οπότε αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα της εντολής σας. Αν συνεργαστείτε με τους στρατιωτικούς δεν θα πετύχετε ποτέ γιατί πάντα θα προσπαθούν να σας κοροϊδέψουν. Θα δούμε, δεν έχει πάει ακόμα εκεί η στρατιωτική δύναμη της ΕΚΟΒΑΣ, δεν έχει πάρει την τελική της μορφή. Αν και η ΕΚΟΒΑΣ έχει καταλάβει αυτό που θέλουμε και τώρα αναφέρεται σε μία ε, δύναμη επιβολής, αν θέλετε, της ειρήνευσης στην περιοχή και όχι μια απλά ειρηνευτικής δύναμης. Πάντως η κρίση δίνει κάποιες ευκαιρίες στη Γουινέα Μπισάου να αντιμετωπίσει επιτέλους το θέμα του εμπορίου ναρκωτικών. Οι γείτονες ε, βλέπουν ότι δεν θα λύσουν ποτέ το πρόβλημα αυτό αν δεν διαγραφεί στη συγκεκριμένη χώρα. Λοιπόν, ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, εδώ ένας πόλεμος μέσω αντιπροσώπων ε, ανάμεσα στην Αγγόλα και την Ιγυρία. Όχι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, αλλά πάρα πολλές διαφορές υπάρχουν στη διεθνή κοινότητα, στην ΕΚΟΒΑ, στα Ηνωμένα Έθνη και νομίζω ότι αν δεν διώξουμε τους στρατιωτικούς θα συνεχίσουν να διοικούν μέσω της διαιρέσεως των υπολείπων. Τώρα για το Σαχέλ, τα σχόλια του κυρίου Τάνοκ. Είναι εκρηκτικό το μνήγμα κύριε Τάνοκ. Υπάρχει κίνδυνος εδώ να καταλήξουμε με μια νέα Σομαλία. Είναι εξίσου έφλεκτο το μείγμα. Έχουμε πάρα πολλές μικρές ομάδες με τοπικές αρμοδιότητες, εξουσίες, εντατικές περιφερειακές αντιθέσεις και πολλοί εξωτερικοί πρωταγωνιστές σε μια περιοχή στην οποία η διακυβέρνηση δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και όπου τώρα υπάρχουν, ε, ε, θα έλεγα, υπάρχει πληθώρα εξοπλισμού στρατιωτικού ε, πολλών τύπων. Τα πράγματα δεν ήταν ποτέ απόλυτα υπό υποέλεγχο, τώρα είναι παντελώς εκτός ελέγχου. Είναι σαφές λοιπόν να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια όλων και της Λιβύης και της Αλγερίας και της Μαυριτανίας και των χωρών Εκοβάσα με την συνεργασία της διεθνούς κοινότητας. Συνεργαζόμαστε επίσης και με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Αφρική και με τις τοπικές χώρες. Μας ανησυχεί ο σύνδεσμος ανάμεσα στην Αλκάιντα Άκμη και το Ιτζιχάντ της Αλγερίας και οι Αλγερινοί ανησυχούν και παίζουν πιο δραστηριό ρόλο για την επίλυση του προβλήματος στο Σαχέλ. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Όσο η κατάσταση παραμένει χωρίς κυβέρνηση τόσο δύσκολο θα είναι να αποκατασταθεί η ηρεμία στην περιοχή για την κατάσταση τώρα στις εξορυκτικές βιομηχανίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς νομοθεσία προετοιμάζεται και σε ποια φάση βρίσκεται η νομοθεσία αυτή. Εμείς είμαστε δραστήριοι όμως στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης εξετάζοντας τα θέματα ακριβώς αυτών των ορυκτών που δημιουργούν σειράξεις ενθαρρύνουμε τους τοπικούς άρχοντες να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία διαφάνειας ITI των βιομηχανιών των επισήμων που προσφέρει περισσότερη ακριβώς διαφάνεια στις δραστηριότητες αυτής της βιομηχανίας. Και όπου επιτρέπεται έτσι να ελέγξουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία <coughs> θα έλεγα είναι καρπός αυτών των δραστηριοτήτων. Για το Σουδάν πάλι, σύντομα. Ένα σχόλιο για το... Για, να, για το κατά πόσο θα δώσουμε μια ευκαιρία στον πόλεμο. Καταρχήν, ε, και οι δύο πλευρές ε, είναι άπειρες ως προς την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Για τον Νότιο Σουδάν ε, η κυριαρχία είναι κάτι καινοφανές και πολύτιμο και θέλουν να την κρατήσουν και να την επιβεβαιώσουν το Βόρειο Σουδάν αισθάνεται μια υπαρξιακή απειλή και ένα κίνδυνο για την ε, διάλυση της χώρας. Οπότε και οι δύο πλευρές ε, αναλαμβάνουν μια θέση επί της αρχής και δείχνουν απρόθυμες και διάλεκτες ως προς το συμβιβασμό. Παρ' όλα αυτά, η πείρα μας δείχνει ότι η χρήση της βίας γενικώ ήταν ένα αποτυχημένο μέσο για επίλυση διαφορών. Και ευελπιστούμε και ότι και οι δύο πλευρές θα το ε, αντιληφθούν αυτό το συντομότερο δυνατό και όσο πιο ομαλά γίνεται και θα επανέλθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Γιατί η κλιμάκωση της βίας θα οξύνει τα προβλήματα και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα λύσει, να τα μετριάσει. Τρεις ακόμη συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ας τους ακούσουμε γιατί από ό,τι ξέρω πρέπει να φύγετε και μετά να ακούσουμε και την απάντηση της κυρίας Μάρσδεν. Το λόγο έχει ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί κάπως από την ανάλυση που έγινε της ε, σύγκρουσης στο Σουδάν. Ομολογώ ότι ήμουν ανέκαθεν ε, της γνώμης ότι αυτή η σύγκρουση είναι μία σύμμετρη σύγκρουση και περισσότερο, περισσότερες ευθύνες εδώ και φτεξίματα έχει η κυβέρνηση του Χαρτούμ. Βέβαια, είμαι υπέρ μια ισορροπημένη θέση προκειμένου να ευοδοθεί, να διευκολυνθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι και πολύ συνεπέ ε, με το σενάριο αυτό να θεωρούμε ότι και οι δύο κυβερνήσει είναι άπειρε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Χαρτούμ είναι άπειρη. Αντίθετα, πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Χαρτούμ ε, έχει πολλά να, παίξει, να κερδίσει υιοθετώντα μια παρελκυστική τακτική που πρόθεσμα θα οδηγήσει στην ανατροπή της κυβέρνησης του Νότου, αν δεν ε, δοθεί μια λύση για το ζήτημα του πετρελαίου. Μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, κατέληξε σε συνενετικό ψήφισμα. Είναι αλήθεια όμως ότι ακόμη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπάρχει μια χώρα, η Κίνα, που επωφελείται από μια παρελκυστική τακτική. Λοιπόν, διαρωτώ η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποια είναι είναι μια θέση περιθωριακή, παρατηρητή, που απλώς ασθενίζεται αυτή την ανάλυση της κατάστασης και ταυτίζεται με μια θέση ανέβρεση ισορροπίας πάση θυσία ή έχει επίγνωση ότι η κρίση μιας ασύμετρης ε, κρίσης ε, θα πρέπει να αναγνωρίσει την ε, φιλοδοξία και της νότιας πλευράς και του νότιου Σουδάν να χτίσει ένα κράτος. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε την προσέγγιση αυτή δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν την επόμενη κατάσταση βρεθούμε πρωτετελεσμένων γεγονότων πολύ πιο επικίνδυνων που δεν θα μας αφήσουν κανένα περιθώριο λιγμό για κάποια επιρροή στο σενάριο αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Mauro. Ευχαριστώ κύριε Μαουρο. Κύριε Λέζινγκ, ευχαριστώ πολύ. Ομολογώ ότι έχω εκπλαγεί από το γεγονός ότι δείχνουν τέτοια έκπληξη συνάδελφοι. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Ντεκεζέρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε, εν πάση περιπτώσει, υποστήριξε και προώθησε την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν, γνωρίζοντας τα προβλήματα και γνωρίζοντας και τι γίνεται με την Αμπέη και τις πλούσιες σε πετρέλαια περιοχές. Τα ξέραμε από την αρχή. Οι σειράξεις ήταν δεδομένες. Και επίση ξέραμε ότι δεν πρόκειται να έχουν λυθεί μέχρι την ανεξαρτησία, ούτε πρόκειται να λυθούν μετά την ανεξαρτησία στο προσεχές μέλλον και το ορατό μέλλον. Με ενοχλεί πάρα πολύ που εκφράζεται τέτοια έκπληξη ε, για τα όσα συμβαίνουν αυτόν τον καιρό. Έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση. Διευκρινιστική και οι περισσότερες. Τι γίνεται λοιπόν τώρα με το σχεδιασμό για μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Τζούμπα. Έχουν προχωρήσει ε, τα σχέδια και ο προγραμματισμός και ποια θα είναι η ακριβής εντολή της αποστολής και το καθήκον. Τι σχεδιάζεται εκεί. Επίσης, υπάρχουν σχέδια των ευρωπαϊκών κρατών να συμμετέχουν στην ενδιάμεση ε, αποστολή στην ΑΜΠΕΗ ε, του Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μουνίθ. Ευχαριστώ. Μάριο Μαουρό, αδίτσο... Ε, κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά ε, μας έθεσε το πρόβλημα κύριος Μαουρό. Το, το ρόλο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κατάσταση στο Σουδάν που την παρακολουθήσαμε από την στιγμή μηδέν και στην οποία θα έπρεπε να κρατήσουμε ένα αποφασιστικό ρόλο και να μην αφήσουμε την κατάσταση αυτή να ε, εγκαταλειφθεί μέσα στις ε, δυναμικές της περιοχής. Ο κύριος Westcott έφυγε δυστυχώς. Μίλησε για τις αιτήσει ε, της ΕΚΟΒΑΣ για κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλιστεί στην υποπεριοχή αυτή μια ασφάλεια. Εγώ θα ε, είμαι κάπω πιο πεζή. Θα ασχοληθώ με πρακτικά θέματα, όχι με τόσο υψηπητή πολιτικά. Γιατί σε λίγο θα ασχοληθούμε και με τον προπολογισμό στην Επιτροπή μα. Ο μηχανισμός σταθερότητας έχει υποστεί σημαντικές περικοπές. Είναι ένας μηχανισμός που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για το πρόβλημα αυτό, μαζί με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, βλέπουμε όμως περικοπές στο μηχανισμό αυτό σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις για τις ανάγκες ε, του επόμενου έτους. Ερωτώ λοιπόν, ε, για να διεκπαιρεώσετε όλες αυτές τις πολιτικές υποστήριξης ευθερότητας της περιοχής που ζητάει η ΕΚΟΒΑΣ και τις αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδότηση ε, της Αφρικανικής Ένωσης έχετε την απαραίτητη πολιτική και οικονομική στήριξη και συμφωνείτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για τον προϋπολογισμό του 2013 και κυρίως για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές έχει προτείνει αισθητές περικοπές στους μηχανισμούς αυτής, ενώ έχουμε ήδη αναλάβει δεσμεύσεις από την Ευρω... ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα έχουμε σημαντικό πολιτικό ρόλο και θα τον στηρίξουμε και με οικονομική παρουσία στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Μουνίθ. Κύριε Μάρτσεν, έχετε ένα πολύ δύσκολο ρόλο τώρα να απαντήσετε στις ερωτήσεις της πολυάριθμης και να καταλήξετε σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις για το Βόρειο και Νότιο Σουδάν. Καταρχήν, πολύ οξυδερκή και προσωπικά και τα σχόλια και εύστοχα της κυρίας Δεκάιζερ, γιατί έχει επιδεινωθεί τόσο η κατάσταση τον τελευταίο καιρό παρά τις προσπάθειες της διεθνού κοινότητα. γιατί πήγαν τόσο στραβά τα πράγματα. Νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που έχουμε να διατυπώσουμε εδώ είναι ότι υπάρχει μια βαθύτατη δυσπιστία εκ μέρους και των δύο κυβερνήσεων. Και δεν είναι περίεργο ότι υπάρχει αυτή η δυσπιστία μετά από δεκαετίες ολόκληρες εμφυλίου πολέμου. Βέβαια θα πρέπει να υποτιμούμε και τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε προσπαθώντας να φέρουμε τις εμπλεκόμενες πλευρές στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και οι δύο κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν την αρχή δύο βιώσιμων κρατών. Στην πράξη βέβαια επανειλημμένως και οι δύο πλευρές υιοθετούν ε, βραχυπρόθεσμες αποφάσεις τακτικής στις διαπραγματεύσεις και δεν υιοθετούν ε, θέση στρατηγικής που να στηρίζει αυτή την αρχή, να ισχύει στην αρχή των δύο βιώσιμων κρατών. Το πάνελ Λεμπέκη είχε πολύ αξιόλογο έργο τους τελευταίους 18 μήνες και έφερε και τις δύο πλευρές ε, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπογραφούν διάφορες συμφωνίες για τη χάραξη των συνόρων, την ορθέτηση των συνόρων, αρχικές συμφωνίες για την ορθέτηση συνόρων, ε, για τους υπηκόους ε, της μιας χώρας στην επικράτεια της άλλης, ε, για το μηχανισμό παρακολούθησης των συνόρων, για την, το MOU για τη μη επίθεση, το μνημόνιο συνεννόησης. Βέβαια, καμία από τις συμφωνίες αυτές δεν έχουν εφαρμοστεί, ούτε καν μερικώς. Απλώς έχουν υπογραφεί. Οπότε, παρερχόμαστε στο θέμα του αν θα έχουν οι δύο κυβερνήσεις την απαραίτητη πολιτική βούληση για να υιοθετήσουν ε, τον ε, δρόμο της ειρήνης και όχι του πολέμου και να προσπαθήσουν να επιλύσουν με ειρηνευτικά μέσα τις διαφορές τους αντί να προσφύγουν στη χρήση στρατιωτικής λύσης ε, ή στρατιωτικής βίας. Και διαρωτόμαστε κατά, πόσο οι δύο κυβερνήσεις χαθούν σε βραχυπρόθεσμα και κοντόφθαλμα τακτικά επιχειρήματα, επιχειρήματα τακτικής, αντί να αναγνωρίσουν την ελεξάρτησή τους και να επενδύσουν στα δύο βιώσιμα κράτη. Στα μέσα Μαρτίου και οι δύο πλευρέ συμφώνησαν ως προς τις διαπραγματεύσεις για το πετρέλαιο ότι θα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ των αξιώσεων του χαρτού και του τι θα μπορούσε η Τζούμπα να πληρώσει στο χαρτούν για να χρησιμοποιεί τον αγωγό πετρελαίου, καθώς και κάποιες μεταβατικές οικονομικές συμφωνίες. Συμφωνήθηκε μετά την πρόταση Εμπέκη ότι οι δύο κυβερνήσεις ε, από κοινού θα ζητούσαν από τη διεθνή κοινότητα να συμβάλλει κατά ένα τρίτο προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το οικονομικό κενό και η Τζούμπα θα αναλάβανε το 1 τρίτο του κόστους, η διεθνής κοινότητα το 1 τρίτο και το χαρτούν το τρίτο τμήμα. Μάλιστα, ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση για επίσκεψη του κ. Μπασίρ στη Τζούμπα, διαπιστώσαμε ότι ήταν απογοητευτική η εξέλιξη παρά την αρχική πρόοδο και είχαμε κλιμάκωση της βίας ε, στα σύνορα και κάποιες συγκρούσεις και εχθροπραξίες μεταξύ των δύο στρατών, των δύο αντιμαχόμενων δυνάμεων. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της Κίνας, έχουμε κοινά συμφέροντα με την Κίνα. Προσπαθούμε να ζητήσουμε από τις δύο κυβερνήσεις να επιλύσουν με ειρηνευτικό τρόπο τα εκρεμή ζητήματα Βέβαια η Κίνα έχει μεγάλη επιρροή στο καρτούν, γιατί έχει στρατηγική εταιρική σχέση με το Χαρτούμ από τα τέλη της δεκαετίας του 80 αλλά έχουν πια οι Κινέζοι σημαντικά συμφέροντα και στο Νότιο Σουδάν και έχει δραστηριοποιηθεί πολύ περισσότερο η Κίνα γιατί οι επιχειρήσεις της ε, άμεσα επηρεάζονται από την σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Εμείς πάντως ε, προσπαθούμε να πείσουμε τις κινέζικες αρχές για συνεργασία και μάλιστα υπάρχει ειδικό Κινέζος απεσταλμένος και στα δύο Σουδάν για να δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε με την Κίνα και να στηρίξουμε το έργο του πάνελ ε, του Εμπέκη. Πιστεύουμε ότι η Διεθνή κοινότητα έκανε ό,τι μπόρεσε για να στηρίξει το έργο αυτού του πάνελ και προσπαθούμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να δώσουμε και πολιτική υποστήριξη στο πάνελ Εμπέκη. Σε ό,τι αφορά την ε, πιθανότητα κατασκευής ε, εναλλακτικού πετρελαγωγού που θα περνάει από την Κένια, η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, είπε ότι θα προτιμούσε καταρχήν ε, να καταλήξει συμφωνία με την κυβέρνηση του Χαρτούν για τη χρήση του πετρελαγωγού. Αρκεί φυσικά η συμφωνία αυτή να έχει λογικούς και δίκαιους όρους και φυσικά ανησυχούν με τις δράσεις ε, της κυβέρνησης του Σουδάν γιατί έχουν δημευθεί κάποιες, ε, κάποια φορτία πετρελαίου και ελπίζουν ε, να αποφευθεί η επανάληψη μιας τέτοιας κατάστασης μετά την συμφωνία με, το Χαρτούμ, με την κυβέρνηση του Χαρτούμ. Πάντως θεωρούμε ότι πιο αξιόπιστη θα ήταν η λύση της κατασκευής εναλλακτικού πετρελαγωγού που θα περνάει από την Κένια ίσως. Είναι σαφές όμως ότι ενώ αρχικά είχαν εξεταστεί και οι πιθανότητες αυτές σε αρχές του έτους. Τελικά όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν δύο με τρία χρόνια για να μην πω πολύ περισσότερο για την κατασκευή ενός τέτοιου πετρελαγού. Οπότε δεν είναι σίγουρο ότι είναι εφικτή και βιώσιμη μια τέτοια λύση. Πάντως η κυβέρνηση του Νότιου Σουδάν εξετάζει πολύ σοβαρά και αυτή την εναλλακτική. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Γνωρίζω ότι για το ΕΚΟ και το Βόρειο και το Νότιο Σουδάν ήταν από τα σημαντικότερα, πιο μεγάλα επίβολα προγράμματα στον κόσμο. Έχουμε φυσικά σημαντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα και στο Νταρφούρ και πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα και στο Νότιο Σουδάν. Αλλά οι ανθρωπιστικέ προκλήσεις στο Νότιο Σουδάν αυξάνονται και διοκώνονται με ρακδαίους ρυθμούς και είχαμε προβλήματα στην πολιτεία Τζόγκλε. Έχουμε πρόσφυγες που φτάνουν στα σύνορα του, του Σουδάν και έχουμε και πρόσφυγες που επιστρέφουν από το βορρά. Οπότε υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα επισητιστικής βοήθειας και ασφάλειας. Οι, ανθρωπιστικ... Οι προκλήσεις πάντως για το ανθρωπιστικό πρόγραμμα είναι τεράστιες και ίσως χρειαστούν περισσότερες ε, ενισχύσεις από τους διεθνείς δωρητές σε ό,τι αφορά το ICC, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την προσχώρηση του Νοτιού Σουδάν στην ε, Συμφωνία του Κοτονού, στην ΑΚΕ, αν τελικά το Νότιο Σουδάν ενταχθεί στο Κοτονού, θα ζητηθεί να υπογραφεί και το καταστατικό της Ρώμης ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ευελπιστούμε ότι το Νότιο Σουδάν θα καταφέρει να ε, τις διαφορές του με το Βόρειο το συντομότερο δυνατό. Σε αυτή κατάσταση και πάλι στο Νότιο Σουδάν για την κυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία και το SPLA, αλλά εν μέρει σχετίζονται με την μετάβαση του Αντάρτικου και τη μετατροπή του σε έναν επαγγελματικό στρατό και ένα αστυνομικό σώμα. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Πάντω χαιρόμαστε για το ότι η κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν αναγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και έδειξε ετοιμότητα ε, και προθυμία να ζητήσει βοήθεια. Νομίζω ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι πολύ θετική. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα τα ζητήματα διακυβέρνηση, η κυβέρνηση Νοτιού Σουδάν έχει προβλέψει, έχει θεσπίσει μια επιτροπή συνταγματικής αναθεώρησης για να επεξεργαστεί το νέο μόνιμο σύνταγμα. Είναι αρκετά περιεκτική η σύνθεση αυτή τη ε, επιτροπή, Περιλαμβάνει και εκπροσώπου ε, μικρών κομμάτων τη αντιπολίτευση. Και μπορεί να επισκιάστηκε το έργο τη επιτροπή αυτή από την κατάσταση στα σύνορα με το Σουδάν. Πάντω η σύσταση αυτή τη ε, επιτροπή Συνταγματική Αναθεώρησης είναι πολύ σημαντική. Και φυσικά συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Νότιο Σουδάν και θα συμβάλλουμε και στην κατάρτιση των δικαστών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο στο Νότιο Σουδάν, η κατάσταση προέκυψε ως εξής ε, εν μέρη. Πέρσι το Δεκέμβριο συνδέθηκε αυτό με τις διαπραγματεύσεις στην Αντίσα Η κυβέρνηση στη Χαρτούμα ανακοίνωσε ότι ε, θα προχωρούσε σε κατάσχεση στο Πορτ Σουδάν ε, κάποιων ε, ποσοτήτων και φορτίων πετρελαίου με τον ισχυρισμό ότι δεν πλήρωσαν τα τέλη που τους αναλογούσαν από τον Ιούλιο, τον Νότιο Σουδάν. Δηλαδή δεν πλήρωσε στο Σουδάν τέλη για τη μεταφορά του πετρελαίου και η κατάσταση επιδεινώθηκε και τέλη Ιανουαρίου, αποφάσισε το Νότιο Σουδάν να σταματήσει εντελώς ε, την παραγωγή πετρελαίου με τον ισχυρισμό ότι η κυβέρνηση στη Χαρτούμ Ε, ε, έπαιρνε από ένα πετρελαγωγό από μια παράκαμψη που είχε φτιάξει ε, πετρέλαιο και το οδηγούσε στα δηληστήρια στη Χαρτούμα αντί να πηγαίνει στο Πόρτ Σουντάν. Σταμάτησαν την παραγωγή εντελώ, την άντληση πετρελαίου. Ήταν πολύ δραστική αυτή η απόφαση. Κανείς δεν την είχε προβλέψει, πιστεύω. Αυτό έκανε όμως τελικά το Νότιο Σουδάν και αυτό είχε προφανώς πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις και πολύ σοβαρές η διεθνή κοινότητα δωρητών Συμπεριλαμβανομένη Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε ε, το Νότιο Σουδάν, δηλαδή να ε, στείλουμε όλα τα κονδύλια που λείπουν από τη χώρα λόγω της ε, διακοπής στην παραγωγή πετρελαίου και είναι μεγάλη ανθρωπιστική πίεση στον πληθυσμό. Η κατάσταση αυτή θα είναι πολύ σοβαρή και τους επόμενους μήνες. Ε, νομίζω ότι έχει διαρρεύσει η έκθεση της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας, θα την έχετε δει κι εσείς. Ε, αυτό δεν αφορά μόνο τον Νότιο Σουδάν και το Σουδάν το ίδιο. Η Χαρτούμ αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη κρίση σε ό,τι αφορά τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και μετά τις επιθέσεις του Νοτιού Σουδάν έχει υποστεί πλήγμα και στα δικά της πετρελαϊκά κοιτάσματα. Είναι ε, πολύ ε, μεγάλο το πρόβλημα της συνοραματικής ε, ισοτιμίας, του πληθωρισμού και έχουν πολύ λίγα συναλλαγματικά αποθέματα. Και το, Σουδάν, και το Νότιο Σουδάν παρακολουθεί τώρα το ένα το άλλο, προσπαθώντας να καταλάβει ποιος από τις δύο χώρες θα καταρρεύσει πρώτος. και αυτό είναι ένα θέμα που επηρεάζει και την πολιτική κατάσταση και τις διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο. Αν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υποστηρίξουμε τον Νότιο Σουδάν, ρωτήσατε. Προσπαθήσαμε από την ανεξαρτησία της χώρας και μετά, συνειδητά, να έχουμε μια ε, ισόρροπη συνολικά ε, αντιμετώπιση. Γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε την εντύπωση στο Σουδάν ότι μετά την ανεξαρτησία του Νότου ρεύουμε την πλάτη μας στο Σουδάν και ασχολούμαστε μόνο με το νότιο Σουδάν. Έχουμε χάσει κάθε ενδιαφέρον μας και εστιάζουμε στο νότο. Ε, καταλαβαίνουμε ότι για τη σταθερότητα του Νοτιού Σουδάν και να είναι η χώρα βιώσιμη είναι απολύτως απαραίτητο. Ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη η ελεξάρτηση με το Βορρά ε, θα πρέπει να υποστηρίξουμε δύο βιώσιμα κράτη και να μην επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο ένα. Αυτή ήταν λοιπόν η υποκείμενη ε, συλλογισμοί στην προσπάθειά μας. Βεβαίως το Νότιο Σουδάν είναι πάρα πολύ φτωχή χώρα και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε και ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και ε, αναπτυξιακή. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που έγινε, ότι πώς, γιατί μας εκπλήσουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Ε, σε σχέση με το ABA και το θέμα του γαλάζιου νήλου ότι δεν είχαν λυθεί αυτά πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδος. Ε, βεβαίως, έχετε απολύτως δίκιο. Διαπιστώσαμε ότι ε, δεν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε ούτε η διαβούλευση ούτε το θέμα της ε, αναδιάταξης των στρατευμάτων των δυνάμεων του SPLA. Και τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση ε, και στο νότιο Κουρτουφάν και στο Γαλαζιονίλο ε, ε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή Αμπέη και θα πρέπει να αποσύρουν τα στρατεύματά τους και οι δύο χώρες όπως θα έπρεπε κανονικά βάσει της συμφωνίας του περασμένου Ιουνίου. Το Νότιο Σουντάν το έχει πράξει και με το νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ελπίζω και η να αποσύρει τα στρατεύματα και να μπορέσει το πάνελ του Πρόεδρου Εμπέκη να αρχίσει να συζητά για το τελικό καθεστώς περιοχής ABA. Κάποιο ρώτησε για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Σουδάν. Υπάρχουν σχέδια και έχουν προχωρήσει πολύ για αποστολή της ΕΠΑΑ που θα εστιαστεί καταρχήν στην ε, βελτίωση της ασφάλειας των αερολιμένα της Τσούβα. Αυτό είναι ένα σχέδιο διακριτικό μεν, αλλά που εξελίσσεται με ταχύ ρυθμού για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ασφάλειας στο αεροδρόμιο της Τζούμπα. Και αυτή θα είναι η ειδική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια τελευταία ερώτηση έγινε για το εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να στείλουν προσωπικό ε, στα, θέματα του ΟΗΕ στην ABA. η αποστολή σε ό,τι αφορά του στρατιωτικού απαρτίζεται αμυγό από θείοπε. Υπάρχουν ορισμένοι πολίτε από άλλε χώρε, αλλά είναι λίγοι σε αριθμό. Και θα μπορούσε να είναι αυτή μια καλή ευκαιρία στα πλαίσια ε, της αποστολής, κοινή αποστολής ελέγχου και παρακολούθησης ε, των συνόρων, να έρθουν και διεθνείς παρατηρητές και ενδεχομένως αυτό θα ήταν μια ευκαιρία ακριβώς για ευρύτερη πλειάδα χωρών και μεταξύ αυτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Μάρστεν. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτού του σημείου της σημερινής διάταξης. One minute break to λεπτού διάλειμμα, παρακαλώ. Το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας και την Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπως και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Αλβανικής Βουλής που ανήκει στην αντιπολίτευση της χώρας για την κατάσταση στην Αλβανία και τη διαδικασία εντάξεως της χώρας. Να καλωσορίσω λοιπόν τους πολιτικούς και άνδρες και γυναίκες από την Αλβανία στην Επιτροπή μας. Παραδοσιακά προσκαλούμε εκπροσώπους της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης γιατί θέλουμε να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος ανάμεσά μας και την Αλβανία αλλά και στο εσωτερικό της Αλβανίας, κάτι το οποίο είναι προϋπόθεση για την λειτουργούσα δημοκρατία να καλέσω τις αλβανικές δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπογραμμίσω τη μεγάλη ανάγκη για την ενίσχυση της δημοκρατίας και την βελτίωση των κοινοβουλευτικών δυνατοτήτων στην χώρα και στην δημιουργία κλίματος πολιτικής ανοχής. Θα θέλαμε επίσης να προχωρήσουν και να καταλήξουν γρήγορα οι διαδικασίες με αποτελεσματικό τρόπο για εκλογικές μεταρρυθμίσεις, θα συνεχίσουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνουμε την Αλβανία να, να συνεχίσει να παίζει ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή, ιδιαίτερα υπό το φως των τελευταίων συμβάντων στην περιοχή, ιδιαίτερα στην Φιρόμ, αλλά και το Κωσυφοπέδιο. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χατζινάστο. Ο κύριος Χατζινάστο λοιπόν. Και αμέσως μετά στους υπόλοιπους ε, Αλβανούς προσκεκριμένους. Θα έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις πολύ θετικές και σημαντικές εξελίξεις που λαμβάνω χώρα στην Αλβανία, καθώς και για την περιφερειακή πολιτική της ε, πατρίδας μου. Εν ώψη της ε, αίτησης της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, βρίσκομαι εδώ μαζί με την κυρία Μπρέγκου, την Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και ε, τον πρόεδρο τη Επιτροπή του Αλβανικού Κοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Θα σε ενημερώσουμε λοιπόν και οι τρει για το πώ έχουν τα πράγματα και θα απαντήσουμε και σε απορίε και ερωτήσει σα. Πρώτα θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εσά προσωπικά κύριε Πρόεδρε για την οργάνωση αυτή τη συνάντηση και να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή σα για την ε, σαφή δέσμευσή τους υπέρ της ε, ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας και της πολιτικής διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Η ενταξιακή διαδικασία είναι πρωταρχική προτεραιότητα για τον αλβανικό λαό. Είναι σημαντικό επίσης ε, εργαλείο για τη διαμόρφωση της ε, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ε, μεταμόρφωσης και αλλαγή της κοινωνίας μας. Έχουμε υπογράψει την πλήρη συμμετοχή μας στην κοινοβουλευτική ζωή και έχουμε ξεκινήσει επικοδομητικό διάλογο με το, Κοινοβούλιο. προσ προσπαθώντας να αποφύγουμε την, να ξεπεράσουμε μάλλον την αποτελμάτωση την πολιτική στην Αλβανία. Ε, ζητήσαμε τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, μας βοηθά επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύουμε όλοι ότι μία πρόοδος ε, προς την εφαρμογή των ε, βασικών προτεραιοτήτων της αγνομοδότησης Επιτροπής του 2010 χρήζουν εθνικής δράσης που ε, στην οποία θα συμμετέχει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό ήταν και το ε, μήνυμα του κυρίου Φίλε, του αρμόδιου επιτρόπου διεύρυνση, ε, στην πρόσφατη επίσκεψή του στα Τύρανα. Σε ό,τι αφορά τι επικείμενε προεδρικέ εκλογέ, όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν διατρανώσει τη δέσμευσή του να εξασφαλίσουν μια εκλογική διαδικασία που θα τηρεί το γράμμα και το πνεύμα του Αλβανικού Συντάγματος η επανάληψη του πολιτικού διαλόγου και τη συνεργασία στο Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδους σημασία για να, συναυθεί, για να σημειωθεί πρόοδος στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια της Αλβανίας. Και μάλιστα οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους κατέληξαν σε ένα σχέδιο εθνικής δράσης και έχουν εφαρμοστεί μέτρα προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος. Η ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 34 ε, τροπολογίες και 27 άρθρα των, ε, του ιστορικού κανονισμού του Κοινοβουλίου και συνεχίζονται οι προσπάθειες για να ενισχυθεί ο ρόλος και το διοικητικό δυναμικό της Βουλής μας ε, για θέματα συναφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλες οι εκκρεμείς νομοθεσίες που ζητούν ειδική πλειοψηφία έχουν εγκριθεί και έχουμε αναλάβει δέσμευση να υιοθετήσουμε και, άλλα, και άλλους νόμους που απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία. Και μάλιστα μία από τις 12 προτεραιότητες που ήταν η θέσπιση του, του γραφείου του διαμεσολαβήτη έχει υλοποιηθεί. Η ad hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος με τη βοήθεια έγκυρων διεθνών εμπειρογνωμόνων ήδη έχει καταλήξει και εγκρίνει πολύ σημαντικέ τροπολογίε που ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του ΑΣΕ και του ΟΝΤΙΡ. Υπάρχει δέσμευση τη επιτροπή να ολοκληρωθεί η εκλογική μεταρρύθμιση εγκαίρως για την προετοιμασία των επόμενων εκλογών. Και η οι βασικέ μεταρρυθμίσει λοιπόν βλέπετε ότι ολοκληρώνονται. Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση τη δημόσια διοίκηση. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε το δημόσιο δίκαιο και να το εφαρμόσουμε πιστά, δημιουργώντα καλύτερη δημόσια διοίκηση. Η στρατηγική τη δικαστική μεταρρύθμιση επίση έχει υιοθετηθεί και ένα σχετικό σχέδιο δράση, καθώ και μηχανισμό παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το σχέδιο αυτό. Προκειμένου να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, έχουμε ήδη μια ειδική επιτροπή που λειτουργεί και η Επιτροπή Νομικής Αρρωγής έχει διευκολύνει την πρόσβαση στην ε, ε, δικαιοσύνη και έχουμε πια ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Έχουμε και ένα νέο εγχειρίδιο για τους ελέγχους που θα χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα βελτιώσει τη λογοδοσία και το δικαστικό κλάδο. Η καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της Αλβανική κυβέρνησης και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στη βελτίωση του νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου καθώς και της ενίσχυσης της θεσμικής συνεργασίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλό πλαίσιο και καλές επιδόσεις στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά η, την κέντρωση, συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων. Καταλήγουμε σε συμβαστικέ λύσει για την άρση ασυλίας υψηλόβαθμων υπαλλήλων και δικαστών. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο επίση είναι ύψιστη προτεραιότητα τη αλβανική κυβέρνηση. Σημαντική πρόοδο έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και τη διοργανική συνεργασία, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, την κατάρτιση τη αστυνομία, καταπολέμηση του ε, λαθρεμπορία ναρκωτικών και διευρυμένη συνεργασία με οργανισμούς και υπηρεσίες εφαρμογής ε, του νόμου. Έχουμε και την στρατηγική για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και προσπαθούμε να βελτιώσουμε το υπάρχον νομικό πλαίσιο. Το Δεκέμβριο του 2011 ε, το, η Διεύθυνση Συντονισμού για τα θέματα ιδιοκτησίας έχει θεσπιστεί και θέλουμε μια σωστή καταγραφή της εκείνης της περιουσίας και σωστές, σωστό σύστημα αποζημίωσης. Έχουμε λοιπόν ένα θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των μειονοτήτων. Οι προσπάθειές μας έχουν στόχο την σωστή εφαρμογή του, ε, του, νομοθετικού, του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Και τον Οκτώβριο του 2011 είχαμε μια απογραφή πληθυσμού με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Το ερωτηματολόγιο της απογραφής περι... περιλάμβαναν ερωτήσεις ε, σε ό,τι φορά την συμμετοχή, τι, ε, ε, την συμμετοχή σε εθνοτικές και φιλετικές κοινότητες με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση προστασία των μειονοτήτων στην Αλβανία με βάση σωστέ στατιστικέ πληροφορίε, Σε ό,τι αφορά την μειοψηφία των Ρωμά, προσπαθήσαμε να, να εφαρμόσουμε τη διεθνή στρατηγική και το, διεθνές, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2010-2015 ε, για την ένταξη, κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Έχουμε, ε, ε, έχουμε μεταφέρει κάποιες αρμοδιότητες από το Υπουργείο Άμυνας στο Υπουργείο Κοινωνικής Ένταξης, προκειμένου κάποιες εκτοπισμένες οικογένειες ε, ε, Ρωμά να ε, βρουν στέγη. Έχουμε επίσης παρεμβάσει σε τομείς σημαντικούς όπως παιδεία και υγεία για να εξασφαλίσουμε πρόσβαση στο Ρωμά και στις υπηρεσίες αυτές. Σημαντικά βήματα έχουν γίνει προκειμένου να αφυπνιστεί το κοινό σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων, να προστατευτούν τα δικαιώματα μου φύλων φιλομεταβατικών, και τα, δικαιώματα των ανηλίκων, των παιδιών και των ατόμων με ειδικέ ανάγκε. Ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ, ένα σχετικό σχέδιο θα περάσει το Μάιο και θα οργανώσουμε και ένα σεμινάριο για την πάταξη τη ομοφιλοφοβία. Αγαπητά μέλη, είμαστε ε, πεπισμένοι ότι σε αυτή την επέτειο της εκατοστής ε, ε, επαιτίου της ανεξαρτησίας μας θα σημειώσουμε σημαντικά βήματα προς την ενταξιακή διαδικασία. Το 2012 είναι μια χρονιά ευκαιρίας για μας και είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με σας για να μετατρέψουμε αυτή την ευκαιρία σε πραγματικότητα. Είχαμε αισθητή πρόοδο σε όλους τους τομείς που σας ανέφερα και παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι έχουμε άλλες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντως έχουμε ένα επικοδομητικό πνεύμα συνεργασία ε, που εφαρμόζεται γενικώ, ώστε όλα τα κόμματα θεωρούν ότι είναι συνυπεύθυνοι ε, αυτή της μεγάλη επιτυχίας ε, της ενταξιακής μας προσπάθειας και έχουμε όλοι αναλάβει δέσμευση για να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ λίγο σε εξελίξει στα Δυτικά Βαλκάνια. Η Ελβανία ενεργά συμμετέχει στην ένταξη της ε, περιοχής και βοηθάει ε, τη συμφιλίωση. Είναι πεποίθησή μας ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης είναι το πιο αποτελεσματικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν όλα τα θέματα του παρελθόντος που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα μεταξύ όλων των κρατών της περιοχής. Είναι επίσης και το καλύτερο αντίδοτο στην αύξηση του εξτρεμισμού που ε, αναδύεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Στις 10 Μαΐου του 2012 ενέκρινε η Βουλή ένα νόμο για τη συνεργασία με τη Γιούλεξ, μια ειδική μονάδα ε, ανάκρισης και έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε πλήρως ε, σε σχέση με ισχυρισμούς ε, που περιέχονται στην έκθεση του ε, γερουσιαστή Dick Marty του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, το 2010. Θα πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα διαπαντός και να αντιμετωπιστούν αυτοί οι ισχυρισμοί. Ενεργά λοιπόν συμμετέχει σε όλε τι περιφερειακέ δραστηριότητε, η Αλβανία που έχουν στόχο να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών, να διευρυνθούν οι περιφερειακές αγορές, να υπάρχει αμοιβαία υποστήριξη για την ένταξη των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Ενεργειακές υποδομές, ε, μεγάλα έργα επίση και άρση κάθε ε, φραγμού επικοινωνίας ε, και ενσωμάτωσης υλικού ΙΑΙΛ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης συνεδριάζει και σε επίπεδο Υπουργό θα συμμετέχουμε ενωμένοι στην πολυμορφία ε, και θα ε, προάγουμε την περιφερειακή συνεργασία. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να καλλιεργούμε τις σχέσεις καλής γειτονίας με τους γειτονές μας για να έρθουμε πιο κοντά όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις σχέσεις με τις χώρες αυτές, καθώς ε, μοιραζόμαστε κοινό μέλλον. Ζουν ε, ο πληθυσμοί αλβανικής καταγωγής σε όλες τις γειτονικέ χώρες και αυτό είναι ε, για μας ένα κίνητρο να προωθηθεί η αιμονική συμβίωση, η ανοχή και η συνεργασία. Στα πλαίσια αυτά η Αλβανία συνεχίζει ε, στη, να συμβάλλει στην ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και έχει και ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον κύριο Μπουσάτη για να μας κάνει τα δικά του σχόλια. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για τον δρόμο της Αλβανίας για την Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργά έχει ενθαρρύνει τη χώρα μου να προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό, σε μεταρρυθμίσεις όπως το πιστεύει και η πλειοψηφία του αλβανικού λαού. Σαν μέλος της αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, θα ήθελα να ανανεώσω το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σε όλους. Η διαδικασία που ακολουθούμε για την ενσωμάτωση της Αλβανίας στις ευρωπαϊκές θεσμικές, ε, στην ευρωπαϊκή θεσμική αρχιτεκτονική είναι κάτι που εμπλέκει το σύνολο των δυνάμεων της χώρας. Θα έπρεπε μέχρι το τέλος του Μαρτίου να έχουμε ολοκληρώσει την εκλογή των ε, εκλογικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούν τα τρία πέμπτα των ψήφων στο Κοινοβούλιο όπως και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την πορεία ένταξης. Βλέποντας την δράση της χώρας από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα, όχι συστηματικά σαν αντοπολιτευόμενος, θα πω ότι η πολιτική συμφωνία του Νοεμβρίου έχει οδηγήσει σε λίγα αποτελέσματα όπως η επιλογή του Ομπούτσμαν με συνενετικό τρόπο και οι νόμοι που απαιτούν για την ψήφισή τους στην πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψήφων. Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η εκλογική μεταρρύθμιση, το κόμμα το κυβερνητικό δεν έχει εφαρμόσει όλες ε, τις ε, αρχές που απαιτείται να ασέβαστη ε, για να υπάρξει εμπιστοσύνη, συνεργασία και αντικειμενική εφαρμογή των εκλογικών ρυθμίσεων. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τα συστήματα επίλυσης εκλογικών διαφορών που θα πρέπει να το σύστημα αυτό να αναθεωρηθεί έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης ε, της ε, σωστής εκλογικής διαδικασίας. Ο στόχος μας είναι να διεξάγονται εκλογές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή στάνταρτς. Αυτό είναι θα έλεγα και συμβολικό σαν κάτι το οποίο θα μας απομακρύνει από τις προηγούμενες εκλογές που ήταν άδικες και ποτέ δεν σεβάστηκαν τα εκλογικά ευρωπαϊκά δεδομένα. Πρέπει λοιπόν πριν ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να έχουμε ολοκληρώσει την εκλογική μεταρρύθμιση. Οι εμπειρίες στις δημοκρατικές κοινωνίες δείχνουν ότι ένα κοινοβούλιο που λειτουργεί πραγματικά εξαρτάται από την εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους. Δυστυχώς όμως οι διαδικασίες αυτές δεν είναι πλέον καθιερωμένες. Ξέρουμε σαν παράδειγμα ότι το να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όταν ο Πρωθυπουργό απευθύνεται φυσικά στον, στο Κοινοβούλιο πρέπει και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης να έχει το αντίστοιχο δικαίωμα. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ισχύει αυτό πάντα τουλάχιστον. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ξεπεραστούν γιατί δυστυχώς επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί το Κοινοβούλιο της χώρας. Πρέπει λοιπόν και η τρίτη προτεραιότητα της Συμφωνίας του Νοεμβρίου, η σωστή λειτουργία της διαδικασίας ψηφοφοριών ε, και της δυνατότητας λήψης του λόγου. Εδώ ε, θα έλεγα οι αποφάσεις ε, του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν έχουν ερμηνευθεί με το σωστό τρόπο. Ελάχιστες από τις αποφάσεις του Προέδρου Τόπη του Μεγάλου Δικαστηρίου έχουν εφαρμοστεί με τον σωστό τρόπο. Αυτά έχουν συνέπειες και για τη λειτουργία του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει οκτώ έδρες και όχι 9 όπως θα έπρεπε και δεν μπορεί να πάρει κατά πλειοψηφία αποφάσεις μερικές φορές. Το ανώτατο δικαστήριο επίσης έχει 16 μέλη και όχι 17 και εκεί δεν μπορεί να υπάρξει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε πλειοψηφία. Ε, φυσικά ε, όλοι λένε ότι θα καλύψουν τα κενά αυτά τις χειρεύουσες θέσεις μετά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτά όλα δείχνουν ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διεξαχθούν σωστά οι εκλογές για τον Πρόεδρο της, ε, η ψηφοφορία μάλλον για την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας. Αυτό θα έλεγα θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι διαφορετικού επίπεδου εξουσίες της χώρας. Όλα αυτά είναι σημαντικά ιδιαίτερα σε τέσσερις τομείς όπου η διεθνής κοινότητα πρέπει να βοηθήσει και έχει ήδη βοηθήσει την Αλβανία στην πορεία για τη δημοκρατία. Επιπλέον, κρίσιμη μάζα ε, συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων είναι πάρα πολύ ουσιαστική για άλλες μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, καταπολέμηση της διαφθοράς, στη δικαιοσύνη, καταπολέμηση ε, του οργανωμένου εγκλήματος, δικαιώματα ε, ιδιοκτησίας, ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους Ρωμά και την άρση των διακρίσεων. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. θα πρέπει να ακολουθήσουμε διεθνείς πρακτικές και πρότυπα για τους ερετούς εκπροσώπους σε ό,τι αφορά τις ασυλίες τους. Και επίσης ε, ε, άλλα σημαντικά νομοθετήματα που χρειάζονται πλειοψηφία τριών πέμπτων και οι ε, μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να ελέγχονται, να παρακολουθούνται, να γίνονται με σωστό τρόπο, με μια ενισχυμένη διοργανική διαθεσμική συνεργασία. Ταυτόχρονα ζητούμε από την κυβέρνηση να συνάδουν τα έργα με τα λόγια τους, γιατί ο χρόνος ε, μετρά αντίστροφα. Θέλουμε να γιορτάσουμε την εκατοστή επέτειο της ανεξαρτησίας μας, ευθυγραμμισμένη με την ευρωπαϊκή προοπτική ε, της ε, χώρας, να προχωρήσουμε στη διαδικασία υποψηφιότητας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση και σας ευχαριστώ για την προσοχή. Κυρία Μπρέγκου, Υπουργό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση τη Αλβανία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι ήταν καιρό πια να μας δείτε όλους μαζί. Όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σας εξηγήσουμε ε, το πνεύμα συνεργασίας, συμπεριλήψης, ε, ενσωμάτωσης όλων. Όλες αυτές είναι νέες έννοιες στην πολιτική μας ζωή από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε εδώ ενώπιον σας, εκπρόσωποι της συμπολίτευσης, της κυβέρνησης δηλαδή, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσωπικά, ε, χαίρομαι εγώ για τη συνεργασία αυτή από τον Νοέμβριο και μετά και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ στενά με τον κύριο Μπουσάτη για να προχωρήσουμε ένα εθνικό ε, σχέδιο και πρόγραμμα δράσης. Ήδη έχουμε συλλέξει τα σχόλια και τις προτάσεις από τη δική του ε, Επιτροπή της Βουλής αλλά και από την Κοινωνία των Πολιτών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή και μεγάλη ευκαιρία για την Αλβανία. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης κύριος Χατζινάστο σας ανέφερε με λεπτομέρειες τις ε, περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ε, προχωρούμε ή ε, επίκυνται το επόμενο διάστημα. Ας πούμε, η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Η αντίστοιχη ομάδα εργασίας προσπαθεί αυτού τον καιρό να μεταφέρει όλες τις προτάσεις που έχουν κάνει και τα δύο κόμματα και έχουν συμφωνήσει παρουσία της ΟΝΤΙΛ και του ΟΑΣΕ Αύριο ολοκληρώνονται τυπικά οι εργασίες, αλλά πιστεύουμε ότι παρόλες τις διαφωνίες που είναι φυσικό να έχουν οι πολιτικές δυνάμεις, θα πριτανεύσει η λογική και ε, ο διάλογος για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και άλλες μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει αυτή η κρίσιμη μάζα, όπως λέμε, για να προχωρήσει η Αλβανία φέτος σε μια νέα φάση, ένα νέο βήμα, θέλετε όχι το καθεστώς υποψήφιας χώρας οριστικά, το οποίο είναι κάτι που χάσαμε ε, δύο χρόνια ε, συναπτά, αλλά θα πρέπει να δείξουμε οριμότητα όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη διαδικασία ε, της ευρωπαϊκής πορείας και να θεωρούμε ότι είναι εθνικό θέμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά για όλους μας. Έχει επέλθει ένα νέο πνεύμα πλέον συνένεσης στην Αλβανία και συνεννόησης και συνεργασίας. Γνωρίζετε ότι πολλοί νόμοι εκκρεμούσαν επί μία διετία στο Κοινοβούλιο. Τώρα ο κατάλογος αυτός έχει εξαντληθεί των νόμων που πρέπει να περνούν με τρία πέμπτα, αλλά ε, επεξεργαζόμαστε ένα νέο εθνικό σχέδιο και κάθε μήνα ε, προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβάλλουμε τις αλλαγές που περνούν από το Κοινοβούλιο ε, σε αυτή την ευρωπαϊκή μας πορεία. Θα ήθελα να ε, δανειστώ ένα από τα μηνύματα που ανέφερε και σωστά ο κύριος Μπουσάτη στην ομιλία του, το θέμα της άρσης ασυλίας. Uh, από το Μάρτιο και μετά στην Επιτροπή Σταθεροποίησης και σύνδεσης έχω πει εξ ονόματος της κυβέρνησης ότι είμαστε όχι απλώς δεσμευμένοι αλλά έχουμε και την προθυμία να ε, θεωρηθεί και νέος όρος για το καθεστώς ε, της υποψήφιας χώρας, το θέμα της ασυλίας. Ε, δεν είναι πολιτικός ο λόγος. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτό στην Αλβανική Βουλή, ότι το θέμα της ασυλίας είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Πιστεύω ότι η άρση της ασυλίας δεν εκφράζεται μόνο, ούτε γίνεται ε, στα λόγια, με ωραία πολιτικά ε, σχήματα, αλλά θα πρέπει να γίνει στην ουσία. Τώρα έχει έρθει η ώρα να γίνει αυτό και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναβληθεί. Το ίδιο ισχύει και για άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι αρκετά σημαντικές από τις 12 ε, βασικές προτεραιότητες ε, που ε, παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη όλοι οι θεσμοί της Αλβανίας και οι εκτελεστικοί οργανισμοί. Όπως σας είπα όμως, Μπορεί μέχρι τον Νοέμβριο να ήταν μεγάλη ανησυχία και την έθεταν όλοι υπόψη μας σε όλες τις ε, συναντήσεις, τις συνεδριάσεις, πάντες εξέφραζαν την ανησυχία τους για την πολιτική κατάσταση στην Αλβανία και μας έλεγαν ότι αν δεν αλλάξει τίποτα μετά τον Νοέμβριο του 2011 ή αν δεν άλλαζε η πολιτική κατάσταση δεν θα προχωρούσε και είμαστε εδώ για να σας αποδείξουμε ότι ο διάλογος που άρχισε ε, συνενετικά τον Νοέμβριο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Και ε, πραγματικά εκεί είναι η διαφορά. Τι δεν συνέβη πριν από μία και τι συμβαίνει σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα και οι υπόλοιπε μεταρρυθμίσεις λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος μπροστά μας και ε, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Παρακαλώ, σας απευθύνουμε όλη η ειλικρινή έκκληση. Προσπαθήστε να μας κρίνετε ε, βάσει του αποτελέσματος και των προόδων. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου αρέσει. Ας προχωρήσουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και να αφήσουμε πίσω μας τις ε, διαμάχες και όσα μας χώριζαν. Ας κοιτάξουμε αυτά που μας ενώνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά και τους τρεις προσκεκλημένους μας από την Αλβανία γιατί μας έκανα μια γενική επισκόπηση της πολιτικής κατάστασης στην Αλβανία και μας διατράνωσαν τη δέσμευσή τους υπέρ της δημοκρατίας, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Θα δώσω πρώτο το λόγο στον κύριο Κούκαν που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Αλβανία και μάλιστα ήταν και ο εμπνευστής της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως ε, για την ευκαιρία αυτή να συναμιλούμε ταυτόχρονα με τους τρεις προσκεκλημένους από την Αλβανία και μάλιστα να βρίσκονται στην ίδια συνεδρίαση και στην ίδια τράπεζα, στο ίδιο πάνελ. Είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η παρουσία. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που λαμβάνουμε κάποιες αισιόδοξε ειδήσει από τα τύρανα. Ε, καιρός ήταν επιτέλους. Γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Επίκυνται προεδρικές εκλογές, επίκυνται η έκθεση προόδου. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά συγκεκριμένα αποτελέσματα από την Αλβανία και χαιρόμαστε ε, για τη δέσμευση όλων των πολιτικών ε, ομάδων και κομμάτων υπέρ του πολιτικού διαλόγου. Είναι πολύ ενθαρρυντική αυτή η δέσμευση και χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι αλλάζει η κατάσταση και αντί να αναλώνεται ενέργεια σε άκαρπες συζητήσεις, φαίνεται ότι αρχίζεται και παιδίδεται στη συνεργασία. Γιατί έτσι θα εντατικοποιηθεί ο πολιτικός διάλογος και θα υλοποιήσετε τις ε, οι δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Αλβανία και τις δεσμεύσεις που θα σας επιτρέψουν να σημειώσετε πρόοδο, γιατί ε, η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος. Χαίρομαι για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ιδιαίτερα του Γενικού Διευθυντή του κ. Σανίνο που πολύ συστηματικά μεταβαίνει στην Αλβανία, στα Τύρανα, έχει συνομιλίες με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο ίδιος ο Επίτροπος Φίλε εκφώνησε πολύ βαρισίμαντη ομιλία ενώπιον της Αλβανικής Βουλής και νομίζω ότι με όλη αυτή την ενέργεια και με τη συνεργασία μεταξύ των αλβανικών φορέων θα έχουμε επιτέλους αυτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι λίγο, αλλά πραγματικά ανυπομονώ. Θε... Περιμένω πολύ πιο γρήγορη πρόοδο από τη χώρα σας. Αύριο θα ακούσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, Υπουργικού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα ακούσουμε και πάλι τη φράση «Όταν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Αλβανίας και όταν υπάρξει αυτή η πρόοδος, μόνο τότε θα προχωρήσει η διαδικασία». Οπότε θα έχετε και ένα επιπλέον έναυσμα. Έχετε την εκατοστή επέτειο της ανάκτησης ανεξαρτησίας της πατρίδας σας και νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να δώσετε στη χώρα σας και στο λαό της να λάβετε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας για την ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται καν να σας επαναλάβω την ε, προθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεργαστεί και να σας βοηθήσει. Νομίζω ότι έχουμε δείξει πολλά και σε αυτή την ε, επιθυμία και την προθυμία. Οπότε το μόνο μήνυμα που έχω να σας μεταφέρω είναι ότι χαιρόμαστε για την αλλαγή που διαβλέπουμε στην Αλβανία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια βελτίωση και την επιδοκιμάζουμε, την επικροτούμε θερμότατα και θα μείνουμε ακόμη πιο υλοποιημένοι αν αυτή η πρόοδος σταθεροποιηθεί και συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κούκαν. Πολύ αισιόδοξη και πολύ θετική αυτή η παρέμβαση. Ο κύριος Χουδής που είναι ο εισηγητής μας για την έκθεση της Αλβανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Αντιπρόεδρο, και Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την Αλβανίδα Πρέσβυρα εδώ, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τους καλωσορίσω στην Επιτροπή μας, να τους ευχαριστήσω για την ενημέρωση που μας έδωσαν για τα βήματα που πράγματι γίνονται, προκειμένου να, πληρώνονται, να πληρωθούν τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους διαβεβαιώσω όπως και ο προηγούμενος συνάδελφος ότι πρόθεσή μας όλου της Επιτροπής και εμένα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να στείλουμε τη χρονιά που η Αλβανία γιορτάζει τα 100 χρόνια της ανεξαρτησίας ένα θετικό μήνυμα, το μήνυμα που περιμένει ο αλβανικός λαός και οι αλβανικές πολιτικές δυνάμεις, να καταφέρουμε να στείλουμε το μήνυμα υπέρ της, του στάτους της ε, υποένταξη χώρας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον τις προόδους και τα βήματα που κάνετε και την προσφορά μας σε ό,τι χρειαστεί να βοηθήσουμε ούτως ώστε να ξεπεραστούν γρήγορα αυτά τα ζητήματα. Επιτρέψτε μου για να κάνουμε και την σημερινή μας συνάντηση, συνάντηση εργασίας για τις μελλοντικές εξελίξεις και μελλοντικές μας εισηγήσεις, να επικεντρωθώ σε δύο-τρία θέματα και θα παρακολούσα Α ε, ε, τον κύριο Αντιπρόεδρο, την κυρία Υπουργό, να μας έδιναν περισσότερες πληροφορίες, αν είναι πρόχειροι, για ορισμένα κρίσιμα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Είναι γεγονός ότι το πολιτικό κλίμα έχει βελτιωθεί, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Η σύνθεση του πάνελ το αποδεικνύει και οι τοποθετήσει σας και όπως είπε και ο κύριος Κούκαν που και αυτός παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, ε, είναι έτσι τα πράγματα. έχετε μπροστά σας τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ε, πείτε μου σας παρακαλώ πώς βλέπετε τις προϋποθέσεις να υπάρξει μια συνενετική λύση για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, πράγμα που δίχως δεύτερη κουβέντα θα βελτιώσει σημαντικά ακόμα περισσότερο το καλό πολιτικό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της Αλβανίας. Το δεύτερο είναι από τα βασικά κριτήρια. Άκουσα τις εξελίξεις που έχετε σχετικά με την υπόθεση της αλλαγής επί το δημοκρατικότερο του εκλογικού νόμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πού καθυστερεί η πλήρη υλοποίηση αυτής της απόφασης, τι δυσκολίες υπάρχουν εδώ, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, πώς να το θέσουμε το θέμα, τι εντοπίζετε εσείς εδώ σε αυτό το, το ζήτημα. Και το τελευταίο, για να μην σας κουράζω, για να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι τον, λόγο, η απογραφή έχει γίνει εδώ, ε, έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα. Τι δυσκολίες έχετε εκεί, τι προβλήματα έχουν προκύψει, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Ε, αυτά θα μπορούσα να σας ρωτήσω και άλλα, όπως καταλαβαίνετε από το ενδιαφέρον, προκειμένου να η έκθεση της Επιτροπής μας να έχει τις καλύτερες δυνατές ε, πληροφορίες, ταυτόχρονα να εντοπίσει σε ποια θέματα πρέπει να ενταθούν ακόμα περισσότερο οι προσπάθειες των αλβανικών δυνάμεων και του αλβανικού λαού, ούτω ώστε πράγματι να γίνει πραγματικότητα στο τέλος, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς που έχει ιδιαίτερη σημασία για σας, να δοθεί θετικό μήνυμα στον αλβανικό λαό, που νομίζω ότι θα διευκολύνει την κατάσταση γενικώ, αλλά ε, μπορεί να βοηθήσει και την ευημερία του αλβανικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή. Ο κύριος Ρότσεκ, που είναι και αυτός ε, πρόεδρος ε, της Ομάδας Εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και να καλωσορίσω τους Αλβανούς φίλους επί σειρά μηνών, για να μην πω ετών, ζητούσαμε τη συνεργασία των ε, βασικών κομμάτων της Αλβανίας. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και τους τρεις και ε, ιδιαίτερα εκπροσώπους και της ε, συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης. Αναφέρατε ότι έχουν επέλθει πολλές αλλαγές στη χώρα από τον Νοέμβριο και μετά. Ναι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής μεταξύ των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων της χώρας και επίσης ως αποτέλεσμα του διαλόγου ε, κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και κοινωνίας των πολιτών. Βλέπουμε αυτή την τεράστια πρόοδο το τελευταίο εξάμεινο. Αναφερθήκατε στις 12 βασικές προτεραιότητες, στο ε, Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης, η ομάδα εργασίας για τις κοινοβουλευτικές μεταρρυθμίσεις, όλες τις μεταρρυθμίσεις που αναφέρεται, το νόμο για τη δημόσια διοίκηση, ε, ε, μεταρρύθμιση δικαιοσύνη, καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Γνωρίζετε λοιπόν ποιε είναι οι βασικές προτεραιότητες. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω δύο-τρία σημεία. Η βασική αδυναμία των τελευταίων δύο-τριών ετών ή ακόμα και πιο παλιά ήταν φυσικά το θέμα των εκλογών. Όποτε γίνονταν εκλογές στην Αλβανία, υπήρχε έδαφος για σύγκρουση. Τώρα τροποποιείται τον εκλογικό νόμο. Γι' αυτό που θα ήθελα να συστήσω ήταν να δεχτείτε τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και της ΟΝΤΙΡ. Γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένας εκλογικός νόμος συνενετικός μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων της Αλβανίας, αλλά κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο σημαντικό οι επόμενες βουλευτικές εκλογές να διεξαχθούν με τρόπο ομαλό και να μπορέσει η διεθνής κοινότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δει πρόοδο απτή και χειροπιαστεί ως προς την εφαρμογή του νεοεκλογικού νόμου. Πριν τις βουλευτικές εκλογές βεβαίως θα γίνουν προεδρικές εκλογές δεν εναπόκειται σε εμά να πούμε ποιο θα πρέπει να εκλεγεί. Αυτό είναι θέμα του αλβανικού λαού προφανώ. Αλλά θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τον συνάδελφο και στι συστάσει για το κλίμα και την ατμόσφαιρα στην Αλβανία. Για περαιτέρω πρόοδο, καλό θα ήταν να εκλέξετε κάποιον που δεν θα είναι διχαστικό. Δεν θα διχάσει την κοινωνία και τη χώρα, αλλά θα την ενώσει. Μίλησε και ο Υπουργό Εξωτερικών για τον περιφερειακό ρόλο της Αλβανίας, που πραγματικά έχει πολύ θετικό ε, μητρό σε αυτά τα θέματα η Αλβανία. Γνωρίζουμε ότι κρεμούν ακόμα κάποια θέματα στα Δυτικά Βαλκάνια και μπορεί η Αλβανία να διαδραματίσει ένα πολύ πρωταγωνιστικό, καταπραγματικό ρόλο σε ό,τι αφορά και τη ΦΥΡΟΜ αλλά και τις διαπραγματεύσεις Πρίστινας Βελιγραδίου ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω ότι η περιφερειακή εξωτερική πολιτική της Αλβανίας θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην πρόοδο. Γιατί η Αλβανία είναι μια χώρα που δεν δημιουργεί προβλήματα και θα πρέπει να αυξήσει το θετικό ρόλο, τον επικοδομητικό που διαδραματίζει στην περιοχή ε, για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ειρήνης στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Με προσέγγισαν κάποιες οργανώσεις παιδιών, που ασχολούνται με παιδιά δηλαδή και ε, διαμαρτύρονται για την κακομεταχείριση παιδιών. Βλέπω μια έκθεση της UNICEF για το 2011 για την κατάσταση των παιδιών στον κόσμο και πραγματικά παραμένουν κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν έχετε προετοιμαστεί να απαντήσετε σε αυτό το θέμα Αλλά θα ήθελα να τονίσω και αυτό το θέμα και να το θέσω υπόψη σας. Δεν ξέρω στις μεταρρυθμίσεις, όταν μιλάτε για μεταρρύθμιση ε, και άρση των διακρίσεων και αυτούς τους νόμους, μην ξεχνάτε τα παιδιά για την κατάσταση ε, των παιδιών στην Αλβανία. Για να μπορούν όλοι να αποφελωθούν από τη βελτίωση της κατάστασης και για το μέλλον των παιδιών, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον της Αλβανίας και της Ευρώπης γενικά. Τέλος, ελπίζω και πάλι ότι αργότερα όταν θα γιορτάσετε την εκατοστή επέτειο της ανεξαρτησίας σας να είναι πολύ θετική η έκθεση πρόοδου και η χώρα σας και με τη δική μας συνεισφορά να προχωρήσει προς το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Ρότσεκ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την αλβανική αντιπροσωπή. Εγώ είμαι Ολλανδός. Στην Ολλανδία υπάρχει μεγάλη συμπάθεια για τη χώρα σας, για το λαό σας και πολλές ΜΚΟ δραστηριοποιούνται. Και από συμπάθεια και από ε, φιλικό ε, πνεύμα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τους πολίτες στη χώρα σας. Ποια είναι η νομική ασφάλεια. Θα πρέπει οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και ε, βλέπω δημοσιεύματα ε, που λέει ότι οι πολίτες στην Αλβανία θα πρέπει να πληρώσουν 90 ευρώ για να φτάσουν στα δικαστήρια. Δεν έχουν πολλοί Αλβανοί 90 ευρώ για να πληρώσουν, για να ε, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στη δικαιοσύνη. Αυτό το θεωρώ σκανδαλώδες. Πέρα από τη λειτουργία της δικαιοσύνης, ποια είναι η δυνατότητα του πολίτη, γιατί αυτό είναι θέμα ε, κράτους δικαίου, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Και κάτι άλλο που ρώτησα και τον Επίτροπο Διεύρυνσης. Ανησυχούν πολύ για τη Βεντέτα. Εκατοντάδες, εκατοντάδες, όχι δεκάδες. Παίρνω γράμματα, εκατοντάδες οικογένειες ανησυχούν. Είναι πάρα πολλοί πολίτες γιατί ε, συνεχίζεται αυτή η ιστορία της Βεντέτας. Τι κάνετε εσείς ως κυβέρνηση, ε, ως κοινοβούλιο για να σταματήσει αυτή η κοινωνική μάστιγα, το έγκλημα αυτό. Μέχρι και η Ολλανδική Εισαγγελία έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πολλοί Αλβανοί δεν ε, μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα σας ε, που ζουν στην Ολλανδία ακριβώς γιατί φοβούνται τη Βεντέτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλτερ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Βιγγένιν. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζινάστη, κυρία Μπρέγκου, κύριε Μπουσάτη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και μας διαμηνήσατε αυτό το πολύ ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα. Κρίμα που δεν ε, έχουμε πολλούς παρόντες για να ακούσουν αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα συνεργασίας από, από την Αλβανία. Και πολλές προσπάθειες έγιναν για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και συνέβαλε σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τρέχουσα κατάσταση στην Αλβανία είναι ο καρπό συντορισμένων προσπαθειών του Κοινοβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά και των, Ευρωπαϊκό, και των Αλβανικών συγγνώμη, οργάνων και φορέων. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, θα έλεγα, ω προ την κατάσταση στην Αλβανία, γιατί θέλουμε σταθερή πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή εκκρεμούν κάποιες σημαντικές αποφάσεις, ε, εκλογικός νόμος, εκλογή του Προέδρου. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί κάποιος υποψήφιος ε, συνενετικός, ώστε η μεγάλη πλειοψηφία του ε, Αλβανικού Κοινοβουλίου να τον στηρίξει. Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, πολύ συχνά ακούμε ότι στο νέο εκλογικό νόμο θα πρέπει να αποφύγεται οπωσδήποτε την επανάληψη της κατάστασης των προηγούμενων περιφερειακών ε, και βουλευτικών εκλογών. Να μην υπάρχουν κενά και παραθυράκια στον εκλογικό νόμο. Προσοχή λοιπόν. Επίσης, πολύ προσεκτικά θα πρέπει να αναλυθεί ο νέος εκλογικός νόμος, αλλά μην καθυστερείτε υπερβολικά την ε, μεταρρύθμιση του. Επισπεύστε παρακαλώ τη διαδικασία για να εγκριθεί ο νέος εκλογικός νόμος το συντομότερο δυνατόν. Μετά τη δέουσα εξέταση όμως. Και μία ερώτηση που δεν σχετίζεται τόσο με την εσωτερική κατάσταση της Αλβανίας, μία ερώτηση προς εσάς κυρία Χατζινάστου. Οι εντάσεις, εθνοτικές εντάσεις της ε, στη Μακεδονία επηρεάζουν, έχουν κάποια απήχηση στην Αλβανία. Ποια είναι η αντανάκλασή τους στην Αλβανία. Και το λέω γιατί αν ρίξετε μια ματιά στην περιοχή, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν ε, κάποιοι θύλακε αστάθεια στα Δυτικά Βαλκάνια και ελπίζω ότι η Αλβανία θα είναι μία από τις χώρες που θα αντισταθμίσει αυτή τη, αυτά τα ρεύματα, τα κύματα αστάθεια, γιατί μπορεί να συμβάλλει στη σταθερότητα και να διαδραματίσει και σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, που είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ιδιαίτερα τώρα και ως προς το Κωσυφοπαίδιο, αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Μακεδονία, λέει ο μιλτής. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιγγένιν. Ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Χρυσόγελος. Ε, Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Μεταξύ των 12 βασικών προτεραιοτήτων δεν αναφέρεται τίποτα για την περιβαλλοντική προστασία πιστεύω ότι θα πρέπει και το περιβάλλον να συμπεριληφθεί ως βασική προτεραιότητα, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά είναι παράγοντας και συνεργασίας ε, εντός της κοινωνίας και μεταξύ των χωρών της περιοχής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην περιβαλλοντική προστασία και στην Αλβανία. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Αυτή ήταν ε, η τελευταία παρέμβαση από τα μέλη της ε, Επιτροπής. Θα ξαναδώσω το λόγο λοιπόν στους προσκεκλημένους μας. Πρώτα στον ε, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα οξιότιμα μέλη που σχολίασαν με τόσο αισιόδοξο, ρεαλιστικό και θετικό τρόπο τις εξελίξεις στη χώρα μου και τις πρόπτικες για περαιτέρω εξελίξεις έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η ένταξη της Αλβανίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για τις ερωτήσεις τις οποίες θέσατε οι οποίες είχαν σαν στόχο το να διευκρινίσουν ορισμένες θετικές εξελίξεις στην διαδικασία της αλβανικής ολοκλήρωσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ και για την αναφορά σας σε ορισμένα θέματα των 12 προτεραιοτήτων του προγράμματος δράσης ουσιαστικά το οποίο έχουμε. Εν πάση περιπτώσει επιτρέψτε μου τώρα να είμαι πιο συγκεκριμένος και να δώσω απαντήσεις. Πρώτον, για τον κύριο Χουντή σχετικά με την εκλογή του Προέδρου. Νομίζω ότι εξέθεσα την άποψη της κυβέρνησης γύρω από το θέμα αυτό. Νομίζω ότι και η κυρία Μπρέγκου και ο κύριος Μπουσάτη ε, έχουν συμφωνήσει εν πολλής. Θεωρείται ότι η διαδικασία αυτή εκλογής θα είναι μια όριμη διαδικασία. Μια διαδικασία η οποία εξακολουθεί να είναι υποδιαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία η οποία σέβεται το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος, ακολουθούνται δηλαδή σαφέστατα οι συνταγματικές προβλεπόμενες διαδικασίες. Μια διαδικασία όμως η οποία δεν αγνοεί όπως είπα και το πνεύμα του συντάγματος. Ο πρόεδρος είναι υπεράνω κομμάτων, ο πρόεδρος πρέπει να είναι σε θέση να αναλαμβάνει σημαντικότατους θεσμικούς ρόλους σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, ε, το δικαστικό, η εξωτερική πολιτική κτλ. Λοιπόν, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Οι συζητήσεις ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα συνεχίζονται ο Πρωθυπουργό πάρα πολύ σύντομα, σαν αρχηγό της πλειοψηφία, ε, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία συζητήσεων ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά σώματα και όπως σας είπα στην αρχή, επανέρχομαι, θα είναι μια όριμη διαδικασία που θα σέβεται το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Τώρα για τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις, τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα υποσυζήτηση θέματα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε και η κυρία Μπρέγκου, συνεδριάζει η Επιτροπή Εκλογικών Αλλαγών ή Μεταρρυθμίσεων. Ασχολείται με τα θέματα που, έχουν, ε, που είναι σε εκκρεμότητα. Θυμίζω ότι το 95% των θεμάτων έχουν διευθετηθεί. υπάρχουν κάποια προβλήματα σχετικά με την κεντρική εκλογική διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν συνεχίζεται και ελπίζω σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε εμείς και το θέμα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής. Δεν περνάω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα σας διαβεβαιώσω όμως ότι υπάρχει διάθεση από όλε τι πλευρέ έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σεβόμενη πλήρω τι βέλτιστε διεθνεί πρακτικέ και σεβόμενη πλήρω φυσικά και τι συστάσει ΟΑΣΕ. Τώρα για την απογραφή, δεν ξέρω τώρα ακριβώς ε, για την απογραφή, πάντως το Σεπτέμβριο θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα της απογραφικής ε, διαδικασίας, η οποία έγινε με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, σεβόμενη ακριβώς τα διεθνή επίπεδα αναφοράς για τις απογραφές του πληθυσμού. Έρχομαι τώρα στον κύριο Ρούτσεκ. Εμείς δεν έχουμε ε, προετοιμαστεί, δεν έχουμε αντιμετωπίσει τα θέματα ε, της κακομεταχείρισης των παιδιών. Πάντως ε, υπάρχουν ορισμένες νομοθετικές διαδικασίες πρόσφατες. Ο νόμος, σαν παράδειγμα, για τα δικαιώματα των ανηλίκων έγινε δεκτός πολύ πρόσφατα και οι εφαρμοστικές διατάξεις για την επόμενη τριετία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή λοιπόν το νομικό πλαίσιο. Το πρώτο Συμβούλιο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών έχει συγκληθεί και θα ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα τα οποία άπτονται της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. για το θέμα της νομικής ασφαλείας και της πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα. Πράγματι, οσδήποτε πολίτης είναι, είναι ελεύθερος να χρησιμοποιήσει το δικαστικό σύστημα και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από το σύστημα αυτό. Δεν γίνεται καμία διάκριση εις βάρος ιουδήποτε πολίτη ή ομάδας πολιτών. Τώρα για τις βεντέτες, τις οικογενειακές ε, αντεκδικήσεις. Αυτά που ακούσαμε σήμερα είναι λίγο υπερβολικά. Έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις τέτοιες. Ε. Έχουν υπάρξει εκκλήσεις για να σταματήσει η διαδικασία αυτή που έχει οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις αιτήσεις, καταθέσεις αιτήσεις χορήγησης ασύλου σε χώρες όπως τη Σουηδία. Ίσως υπάρχουν και κάποιες καταχρηστικές τέτοιες καταστάσεις, περιπτώσεις. Εμείς προσπαθούμε πάντως να ενημερώνουμε τον πληθυσμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης αυτής της διαδικασίας για να ξεκινήσουν μια μεταναστευτική θα έλεγα διαδικασία σε ορισμένες χώρες. Πάντως έχουμε αποτελέσματα, έχουν μειωθεί αυτές οι περιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάται και πολλές φορές όπως είπα είναι περιπτώσεις ε, κατάχρησης ε, του φαινομένου. Το 2011 σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της αλβανικής αστυνομίας είχαμε πέντε περιπτώσεις βεντέτα στην Αλβανία. Πέντε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλοί και δεν ισχύουν αυτά που ακούσαμε εδώ σήμερα. Για τον κύριο Βίγκενιν. σχετικά με το πόσο επηρεάζει η αύξηση των εθνοτικών συγκρούσεων, εντάσεων στην Μακεδονία, λέει ο μιλητής και πόσο επηρεάζουν τη χώρα μου. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε την κατάσταση. Δεν μας αρέσει αυτή η αυξανόμενη η ρητορική σε ορισμένα θέματα, η οποία γίνεται σε, θα έλεγα, σε ένα σκηνικό εθνοτικού τύπου. Νομίζω ότι αυτά τα συμβάντα, αυτές οι ποινικιά κολάσιμες πράξεις πρέπει να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια του νόμου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και δεν θα πρέπει να συνδέονται αυτού του είδους τα φαινόμενα με εθνοτικές εντάσεις. Αυτό προσπαθούμε να πείσουμε ότι πρέπει να γίνει. Οι υπηρεσίες λοιπόν εφαρμογής του νόμου στην χώρα αυτή ε, πρέπει να βασίζονται μόνο ε, στις νομικές ρυθμίσεις που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. Πάντως, στην Αλβανία υπάρχει μια ελάχιστη ρητορική σε σχέση με τα δεδομένα αυτά, με τα συμβάντα αυτά. Από πλευρά ορισμένων μικρών εξοκοινοβουλευτικών κομμάτων γίνονται τα σχόλια αυτά. Αλλά η Αλβανία ως χώρα θεωρεί ότι αυτά τα συμβάντα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη σωστή κλίμακα αντίδρασης και θα πρέπει η κοινωνία της Μακεδονίας, λέω μιλητής, να συνεχίσει την εφαρμογή της πλατφόρμας της Συμφωνίας της Αχρίδας, κάτι το οποίο επιτρέπει ε, την συμφιλίωση και θέτει τα θεμέλια και για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Για το περιβάλλον. Μπορώ να σας πω ότι συνεχίζεται η διαδικασία σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας στο κοινοτικό κεκτημένο και την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας μας σε όλο το κοινοτικό κεκτημένο για τη διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία της φύσης και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτό το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για την Αλβανία. Το περιβάλλον το θεωρούμε κρίσιμο παράγοντα στη μια βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Άρα είναι μόνιμη ανησυχία και μέλημα της αλβανικής κυβέρνησης και αυτό φαίνεται από τη συμπλήρωση της νομικής βάσης για τους τομείς που σας ανέφερα και βεβαίως τα αποτελέσματα είναι καθοδόν. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα επίκυνται, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο, πιστεύω, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ως προς την πολιτική και τα νομικά κείμενα, αλλά και τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Κύριε πρόεδρε της Κυβέρνησης, θέλει κανείς άλλος από τους προσκεκλημένους μας να απαντήσει, να πει μερικά λόγια. Ο κύριος Μπουσάτη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας για τις προτάσεις σας ε, και ε, τις παρατηρήσεις σας ε, σχετικά με την πρόοδο της Αλβανίας προς την Ευρώπη. Δεν είμαι εδώ εγώ για να ερμηνεύω τα λεγόμενά σας, αλλά πώς εκλαμβάνω, ακούγοντας προσεκτικά όλα τα μέλη της Επιτροπής, της απόψας, αναμένεται από την Αλβανία απτά αποτελέσματα, χειροπιαστά, τουλάχιστον αυτά συγκράτησα εγώ ως βασικά σχόλια, μας δίνεται ε, κάποιο περιθώριο χρονικό και περιμένετε σε επόμενες συνεδριάσεις να ομιλούμε όχι στο μέλλον αλλά στο παρελθόν. Να λέμε δηλαδή ποια πράγματα έχουν ήδη υλοποιηθεί και όχι τι πρόκειται να γίνει. Είναι προφανές ότι είναι τέσσερις βασικοί τομείς που χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, δεν θέλω να το παρουσιάσω ως ένα ζήτημα ποσοστού των τροπολογιών και των συζητήσεων που έχουν συζητηθεί και γίνει δεκτές. Το ίδιο ισχύει για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση, γιατί πιστεύω ότι η διαδικασία, η εκλογική και η ενημέρωση και εκπαίδευση ήταν ε, το σημαντικότερο πρόβλημα στις δημοτικές εκλογές και περιφερειακές και κυρίως το θέμα ε, ε, του Δήμου των Τυράννων. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή του Προέδρου και για τη μεταρρύθμιση του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε να λυθούν αυτά μετά από κοινέ προσπάθειες με την πλειοψηφία που είναι στην κυβέρνηση. Ρώτησε ο κύριος Μπέλτερ κάτι για την ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, κρίσιμο και τονίζεται και στην έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως αντιπολίτευση εγώ δεν θέλω να ε, κάνω εδώ πολιτική, αυτό το κάνω στη βόλη της χώρας μου. Αλλά εμείς καταψηφίσαμε το νόμο αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς και πιστεύουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην Αλβανία είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο περίπλοκα από ότι η πρόσβαση αυτή καθ' αυτή. Βεβαίως είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο αυτό και χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και να λυθεί με άλλα νομοθετήματα. που πρόκειται να εγκριθούν και να εφαρμοστούν. Αυτό ήταν το τρίτο. Και το τέταρτο, ζητήματα που έχουν σχέση με τις μεταρρυθμίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την κοινότητα των Ρωμά, την άρση των διακρίσεων, τα άτομα με αναπηρίες. Εδώ θα πρέπει να εργαστούμε και να υποστηρίξουμε πολιτικά την κυβέρνηση ε, για να υλοποιήσει όλες αυτές τις αλλαγές. Έτσι βλέπω εγώ προσωπικά τις εξελίξεις, το προς τα που θα πρέπει να στραφούν έτσι ώστε να έχουμε ε, ένα πιστικό ε, μητρό επιδόσεων ε, για τις 12 βασικές προτεραιότητες που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές για να προχωρήσει η χώρα προς το καθεστώς υποψήφιας. Ευχαριστώ. Thank you Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη χώρα σας και ελπίζουμε οι προεδρικές εκλογές να είναι δίκαιες, δημοκρατικές και σωστές και να γιορτάσετε και ε, ωραία την επέτειο, την εκατοστή της ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας μας διάταξης. Ε, τελευταίο μένο, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί αφορά τα λεφτά. Ε, πρόκειται για την εντολή για τον τριμερή διάλογο ως προς τον προϋπολογισμό του 2013. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τον προπολογισμό του 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει στα τέλη Απριλίου το σχέδιο προπολογισμού και ξεκινάει η διαδικασία του προπολογισμού για το 2013. Στόχο της σημερινής συζήτηση είναι να δώσουμε τη γνώμη μας ότι αφορά τη εντολή του για τον τριμερή διάλογο στις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσουμε το Συμβούλιο. Η γνωμοδότησή μας ε, για τον ε, προϋπολογισμό θα ακολουθήσει σήμερα. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Γιατανμάκη που θα υποβάλει τη γνωμοδότηση ε, στην έκθεση Λαβία που είναι ο κύριος εισηγητής του τμήματος 3 της Επιτροπής Προϋπολογισμών που είναι και η αρμόδια κατουσία. Επιτροπή για την έκθεση αυτή. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Γιατερμάκη, για να μας υποβάλει την γνωμοδότησή της. Θα μιλήσω φιλανδικά. Ευχαριστώ. Γιατί να μην μιλάμε και φιλανδικά, είναι εξίσου σημαντική γλώσσα με τις υπόλοιπες. Θα ήθελα να εκφράσω ε, τη δυσφορία μου σε ό,τι αφορά τη στενότητα του χρονοδιαγράμματός μας. Αλλά η έκθεση του Τζοβάνι Λαβία υπευλή στην Επιτροπή Υπολογισμών την περασμένη εβδομάδα και την περίμενα, περίμενα το σχέδιο έκθεσης ε, για να έχουμε μια βάση για τη συζήτηση και της δικής μου γνωμοδότησης. Εξού λοιπόν και το πολύ πιεσμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε παρά τη βρέχεια προθεσμία. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας μια γενική εικόνα, μερικές πληροφορίες ως προς το υπόβαθρο. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες είναι ριζικά διαφορετική από την κατάσταση που είχαμε πριν από μερικά χρόνια. Απαιτείται εξαιρετική δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα από τα κράτη-μέλη. Είναι χαλεπή κυρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά εφαρμογή αυτής της λιτότητας και της δημοσιονομικής πειθαρχία. Και έχουμε και κάποια παραδείγματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Πολλές είναι οι προκλήσεις του επόμενου προϋπολογισμού, αλλά ίσως ε, αυτοί οι περιορισμοί και οι δυσκολίες μας βγουν σε καλό, γιατί θα μας αναγκάσουν σε κάποιο βαθμό να ξανασκεφτούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, γιατί μια και δεν έχουμε αρκετά χρήματα να κάνουμε τα πάντα, να υλοποιήσουμε όλες τις προτεραιότητες, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ορισμένες από αυτές και να προβούμε σε κάποια ιεράρχηση. Έχουμε πολλές προκλήσεις και στην εξωτερική πολιτική και σε άλλους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν με πολύ προσοχή να εξετάσουμε τις προτεραιότητές μας. Για παράδειγμα, το θέμα της ασφάλειας. Όσο πιο συγκεντρωμένοι είμαστε σε λίγες προτεραιότητες, τόσο μεγαλύτερη ε, επιρροή και βάρος θα έχουμε στη συζήτηση. Πάντως, καθήκον της δικής μας Επιτροπής είναι να στείλει ηχηρά πολιτικά μηνύματα και να συμβάλλει στην ανέβρεση των σωστών λύσεων για τον προϋπολογισμό. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ίσως αυτή τη φορά κληθούμε να κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εξαιτίας, επαναλαμβάνω της ε, δύσκολης οικονομικής μας κατάστασης. Όλοι ξέρουμε ότι οι εξωτερικές υποθέσεις δεν είναι η ύψη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και το πιο προσφυλές θέμα σε όλους. Πάντως και η δική μας Επιτροπή και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, έχει ένα ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα μπούμε και σε ένα νέο πολύ σημαντικό σε ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είμαι βέβαια όμως ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα κριτήρια του προϋπολογισμού. Έχουμε προβλήματα και με την ανάπτυξη που χωλαίνει και αυτή. Και θα πρέπει να διαρωτηθούμε πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις. Έχουμε κάποια θέματα που είναι ευαίσθητα, μεν, αλλά θα πρέπει να διαρωτηθούμε για παράδειγμα τι γίνεται με την διεγκόμενη κάθε χρόνο ε, οικονομική ενίσχυση προς την Τουρκία ενώ η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας ε, είναι γύρω από το 10% και η οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης είναι πολύ χαμηλότερη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι 10%. Και μάλιστα σε μερικές χώρες δεν είναι καν θετική η οικονομική ανάπτυξη. Έχει θετικό πρόσημο μόνο σε λίγες χώρες μέλη. Ενώ η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας είναι σαφώς ε, μεγάλη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται και μάλιστα ενισχύεται η οικονομική ενίσχυση προς τη χώρα αυτή. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια του προϋπολογισμού. Οι απλοί πολίτες, ε, ακόμη και μερικοί ευρωβουλευτές, ε, δεν μπορούν ε, να κατανοήσουν με σαφήνεια πώς δαπανώνται τα κονδύλια της εξωτερικής πολιτικής. Οπότε δεν μπορούμε να δούμε και τι αξιοποίηση γίνεται αυτών των κονδυλίων, τι αντίκτυπο έχουν και κατά πόσο πιάνουν τόπο. Και ακόμη ε, όταν ξέρουμε πού πηγαίνουν τα κονδύλια δεν είμαστε βέβαιοι για το αν αξιοποιούνται σωστά και τι αποτέλεσμα έχουν. Αν δείτε κανείς τι κάνει στον οικοκυριό του, διαπιστώνεται ότι ο καθένας ξέρει πού πάνε τα λεφτά του. Εδώ έχουμε όμως δημόσια κονδύλια, έχουμε κονδύλια των φορολογουμένων, τα χρήματα των φορολογουμένων και φαίνεται να μην μεριμνούμε για την παρακολούθηση της πορείας τους μέχρι την χρησιμοποίηση και την αξιοποίησή τους. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε μια διαφάνεια στη διαδικασία του προϋπολογισμού για να γίνει όσο πιο ανοιχτή γίνεται. Και σε, ό,τι αφορά τα αποθεματικά μας, άλλο σημαντικό θέμα. Θα πρέπει και αυτό να το προσέξουμε μαζί με τον τρόπο αξιοποίηση των κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την οργάνωση του προπολογισμού μας. Κάτι που δεν είναι απλό. Και θα πρέπει να διευκολύνουμε φυσικά τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά, αυτή είναι μια σύντομη εισαγωγή. Είμαι όλη αυτά, αυτιά τώρα, περιμένω τα σχόλια των μελών της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάκη. Συγγνώμη που δεν είπα προηγουμένως σωστά το όνομά σας. Και τώρα οι σκιώδες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κύριος Μιχαήλ Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ε, ε, στα φιλανδικά ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Γιατενμάκη, η ε, αγαπητή Άνελη, όλες οι γλώσσες βεβαίως είναι ίσες, γι' αυτό στα λέω αυτά φιλανδικά και γίνω στα γερμανικά τώρα. Σας ευχαριστώ για τις σκέψεις, τις προτάσεις ε, της συναδέλφου. Είναι γεγονό ότι όπως έχει κατάσταση σήμερα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ε, έχουμε δαπάνες ε, που θα αποδειχθούν στα μάτια της κοινή γνώμης άσκοπες, περιτές ή σπατάλες. Θα πρέπει πάντα να είμαστε πολύ στοχευμένοι, πολύ προσεκτικοί και πολύ φιδωλοί στη διαχείριση των χρημάτων μας για να πιάνουν όσο γίνεται περισσότερο τόπο. Αυτό είναι αναμφίβολο και δεν το αμφισβητεί κανείς. Εδώ συμμετέχω πολλά χρόνια εγώ στο Κοινοβούλιο και στην πρακτική εφαρμογή της εξωτερικής μας πολιτικής ανέκαθεν μιλούσαμε για χρόνια υποχρηματοδότηση και σωστά την καταγγέλαμε αυτή. Διότι αυτό που μας χρειάζεται είναι να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο, ένα ενεργό για να είμαστε μια ένωση που να έχει σημασία, να έχει παρουσία και να μπορεί να ε, υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να διαθέτουμε και τα ανάλογα κονδύλια. Το πρόβλημα με την εξωτερική πολιτική είναι το εξή. Σε αντίθεση με τα επταετή προγράμματα για τα διορθωτικά ταμεία, για τον πολιτισμό ή για άλλε πολιτικέ μα, στην εξωτερική πολιτική μπορεί να συμβεί κάτι τελείω απρόπτο από τη μια μέρα στην άλλη και δεν μπορεί να το προγραμματίσει. Ούτε θεομηνία προγραμματίζεται, ούτε πόλεμο, ούτε οι επιπτώσει που μπορεί να έχει μια σύραξη η διάρκεια που μπορεί να έχει μια σύραξη. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Και θα σας παρακαλούσα στη διατύπωση να επιλέγαμε ένα τρόπο, στα αγγλικά ας πούμε, επαναλαμβάνει για να επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, ότι θα πρέπει να προβλέπονται επαρκή κονδύλια στον κοινοτικό προπολογισμό. Όλα αυτά τα διάβασα αγγλικά. Είναι σημαντικό να πούμε λοιπόν σε σχέση με αυτό ότι ισχύει κάτι τέτοιο στην εξωτερική πολιτική. Και όταν έχουμε περικοπές, να μην εγκάρσει σε γενική προσπάθεια αλλά στοχευμένη προσέγγιση σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού. Στοχευμένη όμως συνειδητή και όχι γενικά και αόριστα σε όλα τα κονδύλια. Άλλο. Συμφωνώ να υποστηρίξουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν προγράμματα που δεν εφαρμόζονται ε, ικανοποιητικά και θα πρέπει να εγκαταλείπονται. Είναι σωστό όμω και σημαντικό να μας τα εξηγεί αυτά επαρκώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το αξιολογούμε εμείς και να ε, καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Σε ό,τι αφορά το σημείο 3, είναι σημαντικό πιστεύω και εκεί και στην Ανατολική γειτονία και στην Νότια γειτονία να κάνουμε τα δέοντα. Και ποια είναι τα δέοντα. Και στις δύο περιφέρειες χρειάζεται να γίνουν πολλά, γι' αυτό θα πρέπει και στις δύο να γίνεται ρητή αναφορά. Και έχω μια ερώτηση προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περικοπές στην νότια γειτονία της τάξης του 3%. Ε, μήπως είναι λάθος μήνυμα αυτό. Λέμε για την, την ε, Αραβική Άνοιξη ότι μπορεί να έχει αποτύχει σε κάποιες χώρες ή να έχει λοξοδρομήσει σε κάποιες άλλες. Και τώρα μειώνοντας τον προπολογισμό εμείς βοηθούμε αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή να δώσουμε την εντύπωση ότι δεν συμφωνούμε ας πούμε, με την κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγματα και οι εξελίξεις στις αραβικές χώρες. Προσοχή μεγάλη χρειάζεται εκεί και να επενδύσουμε πολλά ακριβώ για να στραφούν τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά με ενδιαφέρει αυτές οι δύο γεωγραφικές περιοχές να έχουν ισόρροπη αντιμετώπιση και να αναφέρονται ρητά και η Ανατολική Γειτονία και η Νότια. Στο σημείο 4 τώρα. Πολύ συχνά έχω ζήσει τέτοιε καταστάσει Να είναι πολύ λίγα τα κονδύλια και μετά να αυξάνονται με τροποποιητικές ε, επιστολές. Παράδειγμα Παλαιστίνη. Αυτό θα πρότεινα μια άλλη διατύπωση ε, καλή μια δέσμευση δαπανών που θα αντανακλά τις πραγματικές ανάγκες από την αρχή του οικονομικού έτους για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει ε, σωστά αυτές τις προσπάθειες. Κάπως έτσι να είναι η διατύπωση στα αγγλικά. Στο σημείο 5 εγώ θα το διήβρινα. Δεν είναι μόνο το θέμα της αρκτικής και της βόρειο-ευρωπαϊκής διάστασης. Εγώ είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό. Ε, είναι η ευρύτερη περιφέρεια ευρωπαϊκή. Δεν είναι μόνο η βόρεια διάσταση. Ε, Στο σημείο 6 είναι σημαντικό να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της Ένωσης και την ε, προβολή προς όλους. Αυτές ήταν οι πρώτες παρατηρήσεις για το κείμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Gala. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Βουίλης. Ο κυρία Μουνή, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εγώ έμεινα ευρώντη από την γνωμοδότηση που μας παρουσίασε η κυρία Γιατερμάκη που συμμετείχε και πέρυσι στην ε, αντιπροσωπεία στον τριμερή διάλογο. Όλοι συμφωνούμε υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά δημοσιονομική πειθαρχία δεν σημαίνει κατά ανάγκη να θυσιάσουμε τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, γίνουν σε, να είναι σε παγκόσμιο προσκήνιο σημαντικός παράγοντας. Φαίνεται όμως ότι φέτος έχουμε μια γνωμοδότηση που θα μεταβιβάσουμε στην ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού που θα συμμετέχει στο τρι... στον τριμερή διάλογο που έρχεται σε αντίφαση με τη γραμμή που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια και που μας υπενθύμισε ο κύριος Γκάλερ. Δηλαδή το τμήμα 4 κα... κατά παράδοση υποχρηματοδοτείται. Ενώ αν θέλουμε μια πραγματική αποτελεσματική πολιτική, εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίσουμε και επαρκή χρηματοδότηση. Διαφάνεια. Φυσικά και είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Το ανέφερε αυτό η κυρία Γιαταρμάκη. Αλλά διαφάνεια από μόνη τη δεν σημαίνει λιγότερα κονδύλια, αλλά καλύτερη αξιοποίηση και καλύτερη ενημέρωση για τον τρόπο αξιοποίηση, όχι περικοπή των κονδυλίων. Επίσης, δεν μπορούμε να λέμε ότι θα πρέπει ε, να προβούμε σε περικοπές γιατί ε, διανύουμε εποχή λιτότητας. Το θέμα είναι πού θα κάνουμε τις περικοπές ώστε να μην ε, παραβλάψουμε τις εύλογες φιλοδοξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν σημαντικός διεθνής παράγοντας. Επίσης, δεν μπορούμε να λέμε ότι διαφωνούμε ή μάλλον ότι συμφωνούμε με τις περικοπές των κονδυλίων σε προγράμματα που δεν εκτελέστηκαν σωστά. Αυτό όμως δεν θα μπορεί να μεταφράσει σε οριζόντια περικοπή όλων των προγραμμάτων. Θα πρέπει να δούμε ποια προγράμματα δεν λειτουργήσαν σωστά και σε αυτά να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Και όχι οριζόντια να γίνουν περικοπές σε όλα τα προγράμματα. Διαφωνούμε με αυτή την ανετιολόγητη οριζόντια περικοπή σε πολλές δημοσιονομικές γραμμές αυτών των προγραμμάτων. Ένα άλλο σημείο που επίσης είναι ανησυχητικό είναι εκεί που αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σημείο 2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει τεχνητά διωγγώνει ορισμένες προτάσεις της κατηγορίας 4 για να διευκολύνει τη συνδιαλλαγή και την συζήτηση στον τριμερή διάλογο. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια χρηματοδότηση είναι γιατί έχει υπολογίσει τις ανάγκες της, όχι για να διευκολύνει τη διαπραγματευτική της θέση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κατά παράδοση ζητούμε διόρθωση της υποχρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας του τμήματος 4. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι ε, η επαρκής χρηματοδότηση γίνεται μόνο και μόνο για τη διευκόλυνση της διαπραγματευτικής ισχύω της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Γκάνερ για το σημείο 5. Σημαντικές είναι η αρκτική και η βόρεια διάσταση. Αλλά αν αναφέρουμε αυτές τις δύο διαστάσεις, αναφέρουμε και τις άλλες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής ένωσης που είναι εισάξιες. Και το είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ε, πολιτική γειτονία με τον Νότο, για παράδειγμα, είναι σημαντική. Η πολιτική με τη Λατινική Αμερική, που συνδυάζεται και με την Επιτροπή, τη Στρατηγική 2020. Και αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην εγγραμμοδότηση. Να αναφέρονται επίση και άλλε διαστάσει που είναι σημαντικοί άξονε τη εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλο, ό,τι αφορά το σημείο 4 τη ΟΝΡΑ και τη χρηματοδότηση τη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκάλερ να διορθώσουμε τη διατύπωση Θεωρώ η γνωμοδότηση της κυρίας Γιατεμάκη, την οποία ευχαριστώ εμπαρόδο για το έργο της, γιατί άσχετα με τα αποτελέσματα το έργο πρέπει να αναγνωρίζεται, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να επανατοποθετηθεί με τελείως διαφορετικούς όρους αντίθετους, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ στο τριμερή διάλογο ή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σωστή η έκθεση του Γενικού Εισηγητή του κυρίου Λαβία από, ως προς τις απαιτήσεις της δικής μας Επιτροπής, από ότι η ίδια γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής που είναι η γνωμοδότηση της κυρίας Γιατανμάκη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μουνής για τους πρασίνους τώρα. Κυρία Μπραντνερ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για το κείμενο. Έχω κυρίως ερωτήσεις εγώ να κάνω. Στην πρώτη παράγραφο λέτε ότι δεν θα πρέπει να εξαιρεθεί από τις περικοπές και αυτός ο προϋπολογισμός. Θα πρέπει όμως να λέτε και πού θα γίνουν οι περικοπές. Και εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Να πούμε εδώ θα περικόψουμε, δεν ξέρω πού, Λατινική Αμερική ή αλλού, αλλά να λέμε γενικά περικοπές χωρίς να δίνουμε κάποια κατεύθυνση, ε, το θεωρώ δύσκολο. Γι' αυτό ρωτώ κυρία Γιατιμάκη, τι έχετε υπόψη σας. Θα μπορούσατε να το συγκεκριμενοποιήσετε για να συμφωνήσω. Γενικά και αόριστα δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω. Στη δεύτερη παράγραφη συμφωνώ και θέλω να ρωτήσω και εγώ το ίδιο με την κυρία Μουνίθ. Πού είναι η τεχνητή αύξηση. Τουλάχιστον να το συγκεκριμενοποιήσετε, να το ορίσετε. Πού έχουμε τεχνητή αύξηση της χρηματοδότησης. Το συγκεκριμενοποιήσουμε ξανά. Γιατί αλλιώς θα ζητήσω απόρριψη. Στο σημείο 3 έχω την εξής ερώτηση. Ε, ε, ε, κάτι σημειώνεται και καλωσορίζεται κάτι για την Ανατολική γειτονία, για τον Νότο τίποτα. Μετά τις δραματικές αλλαγές που γίνονται στην Νότια όχθη της Μεσογείου, με εκπλήσει αυτή η αναφορά. Αν μη τι άλλο, αναφέρετε την Ανατολική γειτονία, να πείτε κάτι αντίστοιχο και για την νότια γειτονία. Υπάρχει πολιτικός λόγος που την έχετε παραλείψει. Για ποιο λόγο δεν αναφέρετε καθόλου τον Νότο και μόνο την Ανατολή. Άλλες ερωτήσεις. για την υποχρηματοδότηση και στην πολιτική γειτονία. Ακριβώς δεν έχουμε αρκετά χρήματα. Και κάτι που μου λείπει από την έκθεση. Ε, πιο συγκεκριμένα πόσο μας κοστίζει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης. Αναφέρεστε σε ποσοστά 5,7%. Από πού όμως προέρχεται αυτή η αύξηση. Έχετε θέσεις ε, άντε 14. Από 108 αυξάνονται αυτές οι θέσεις σε 119. Γιατί χρειαζόμαστε τόσο υψηλό βαθμός και μάλιστα 11 του χρόνου ε, σε ε, βαθμό άντε 14. Πώς μας προέκυψε αυτό. Άλλο θέμα, πάλι για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Κάτι που με εκπλήσει πολύ είναι η αύξηση στον προϋπολογισμό των υπηρεσιών ασφαλείας στις εξωτερικές μας ε, αντιπροσωπείες. Αυξήθηκε αυτό κατά 30 περίπου της 100 και ρωτώ πώς έγινε αυτό. Και σε ποιες χώρες αυξήθηκε τόσο πολύ η ασφάλεια, τι συμβάσεις είναι αυτές. Κάτι άλλο που θέλω να καλωσορίσω είναι τα χρήματα στο πιλωτικό πρόγραμμα που είχαμε για μια διετία για την πρόληψη ε, των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση. Αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα μπήκε ως κανονική πίστοση στον προϋπολογισμό και χαίρομαι γι' αυτό ε, και θεωρώ σωστή την αύξηση της πρικοδότησης επίσης. Θα σας παρακαλούσα να μου διευκρινίσετε τις ερωτήσεις που σας έκανα για να κάνουμε αντίστοιχα και τροπολογίες. Για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστούμε κυρία Μπραντνερ. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Γετερμάκη, για να σχολιάσει αν θέλει τις απόψεις των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις, πάρα πολύ εύστοχες. Είμαι σίγουρη ότι σε μελλοντικές συζητήσεις θα μας απασχολήσουν ξανά. Θα ήθελα να πω μόνο ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλω να απομακρυνθώ από το παγκόσμιο ρόλο της Ένωσης. Τι είναι όμως σήμερα ο παγκόσμιος ρόλος που διαδραματίζει η Ένωση. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αν θέλουμε να επικεντρωθούμε κάπου. Άρβοα. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μία γεωγραφική περιοχή, μπορεί να έχει μεγαλύτερη επιρροή η Ένωση γενικότερα. Το γεγονός ότι αυξάνονται οι δαπάνες δεν σημαίνει ότι πιάνουν και τόπο. Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Είναι συνθήκη ικανή, αλλά όχι αναγκαία. Και αυτό δεν είναι θέμα του προπολογισμού και μόνο, γενικά θα πρέπει να μα απασχολήσει ποιο είναι ο παγκόσμιος ρόλος της Ευρωπαϊκής. Μειώνεται συνεχώ ο ρόλο μα και πώ θέλουμε να χρησιμοποιούμε σωστά πλέον τους ε, λίγου οικονομικού πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα. Πού πρέπει να γίνουν οι περικοπές, ρωτάτε. Αυτό είναι μια κοινή απόφαση Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται η Αραβική Άνοιξη δεν σημαίνει περικοπές στη γειτονία προς Νότον, αφού ρητά αναφέρθηκα εγώ στους Παλαιστινίου, για παράδειγμα. Συμφωνούμε όμως όλοι ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει παρουσία και επιρροή. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στην Αραβική Άνοιξη. Ρωτήσατε για την αύξηση των δαπανών στις υπηρεσίες ασφαλείας. Αυτό μάλλον απευθύνεται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο και για τα πιλωτικά προγράμματα. η Την αποφυγή συγκρούσεων και την πρόληψη. Δεν υπάρχουν σημεία που θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να αυξήσει την επιρροή της. Νομίζω καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθούμε στην άμεση γειτονία μας και να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιατερμάκη. Να σας δώσω για κάποιες πληροφορίες ε, για την προθεσμία για τις τροπολογίες που λύγει αύριο, 15 Μαΐου, 12 το μεσημέρι και θα πρέπει να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά γιατί ο χρόνος πιέζει. Επόμενη συνεδρίαση αύριο 15 Μαΐου 5 με 6 και 4 με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Λιβύης για την τρέχουσα κατάσταση και τις επερχόμενες εκλογές. Η κυρία Μουνής, τι θέλετε. Ένα διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ για την απουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, ΑΕΔ, γιατί συνήθως όταν εξετάζουμε τον προϋπολογισμό, καλό θα ήταν να έρχεται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σχολιάζει τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία διαμαρτυρία λοιπόν για αυτή την απουσία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για τις τροπολογίες. Ακόμη δεν έχουμε λάβει τα έντυπα τα, τυποποιημένα για την υποβολή των τροπολογιών. Παρόλο που είπατε ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι λίγη προθεσμία. Και επίσης μετά τις απαντήσεις κυρίας για την Μάκη θα ήθελα να σχολιάσω ως προς το περιεχόμενο ότι το 2011 το Ισραήλ κατέστρεψε 59 έργα που είχε χρηματοδοτήσει την Παλαιστίνη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην μειώσουμε εκεί τα κονδύλια αντί να περιορίσουμε την ασφάλεια στην ΙΕΔ και γιατί να μην ενισχύσουμε την ειρηνευτική διαδικασία και τα μέτρα ασφάλειας αλλού. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο και για τη συζήτηση και για την αποσαφήνιση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Όταν αναθέτουμε την σύνταξη γνωμοδότηση σε κάποιον, δεν θα πρέπει να εκφέρει με αυτή προσωπικέ του απόψει, αλλά να εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα απόψεων τη Επιτροπή. Ευχαριστώ μία διευκρίνηση. Ίσως δεν καταλάβατε. Αύριο λίγη η, ε, η προθεσμία, όχι για την γνωμοδότηση της Επιτροπής που θα δώσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά για την εντολή ως προς τον τριμερή διάλογο. Δεν τροποποιούμε τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό, μόνο ε, για την εντολή του τριμερούς διαλόγου ισχύει η αυριανή προθεσμία. Πάντως, όντως, κυρία Μονής, την περασμένη Τετάρτη ε, λάβαμε το έγγραφο και ούτε μια εβδομάδα δεν ολοκληρώνεται μέχρι αύριο. Όντως είναι πολύ σύντομος ο χρόνος. I was uh, advised by our at that η Γραμματεία με ενημερώνει ότι θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου, όπως και άλλες επιτροπές. Οπότε όντως δεν έχει μείνει και πολλής χρόνος για την κατάθεση τροπολογιών. Can I say very realistically, we won't... Δεν θα διαπραγματευτούμε την Πέμπτη Παρασκευή από ό,τι φαίνεται, αλλά με του κοιόδη ηγητέ ε, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν έχει νόημα. Είτε αύριο είτε την Τετάρτη λήξη προθεσμία το ίδιο είναι. Για μας δεν έχει διαφορά. Okay, I leave this uh, uh, to... Can we agree on Wednesday? So we agree on one... Να συμφωνήσουμε και την Τετάρτη, καλώς. Εντάξει, Τετάρτη μεσημέρι τότε. Τετάρτη μεσημέρι λίγη προθεσμία. Τελευταίο σημείο ήταν αυτό στην ημερήσια διάταξη. Καλό σας απόγευμα και ραντεβού αύριο.